Sechs. Morgen, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Erster Tagesordnungspunkt. Καλημέρα σας. Στο πρώτο σημείο της σημερινής διάταξης σήμερα έχουμε την ε, μελέτη αντικτύπου και έχουμε τον κύριο Τσίστερα, ο οποίος είναι ο εισηγητής. Έχετε το λόγο, κύριε εισηγητά. Well, Chairman, thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαστε τόσο πολύ άριθμοι συνάδελφοι στην αίθουσα για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μπαίνω στον πειρασμό να μακρηγορήσω όλα ώστε να έχουν και άλλοι συνάδελφοι την ευκαιρία να καταθάσουν. Είχαμε πολύ χρήσιμη συζήτηση για την γνωμοδότηση αυτή, κυρία Πρόεδρε, όταν δεν είχε ακόμη αποκρισταλωθεί, ήταν ακόμη σχέδιο πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά η θέση δεν έχει αλλάξει έκτοτε. Οπότε ουσιαστικά περιμένω τις προτάσεις και τις τροπολογίες των συναδέλφων πριν περάσουμε σε πιο διεξοδική συζήτηση. Πάντω ε, ανακεφαλαιώνω. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση σε μια έκθεση πρωτοβουλίας για τα, τις μελέτες επιπτώσεων και την προσπάθεια ανεξαρτητοποίηση αυτών των μελετών. Εγώ είμαι υπέρ τη ανεξαρτησίας αυτών των εκτιμήσεων του αντικτύπου. Όταν ενισχύσουμε την ανεξαρτησία τους θα τους προσδώσουμε και περισσότερη αξιοπιστία. Στη γνωμοδότησή μου κάνω διάφορες προτάσεις για το πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτή η ανεξαρτησία. Ίσως η πιο δύσκολη πρόταση, πιο δυσεφάρμοστη, είναι όταν τροποποιείται μια νομοθετική πρόταση από το πέρασμά της σε μια επιτροπή, σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή, η μελέτη επιπτώσεων να εξυγχρονίζεται, να επικαιροποιείται υπό το φως των ε, τροπολογιών που έχουν ε, εγκριθεί και των αλλαγών που έχουν γίνει σε μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Βέβαια, αυτό είναι αρκετά δυσχερές, ε, δεδομένου του στενού χρονοδιαγράμματος που ισχύει πολλές φορές. Πάντως, αν θέλουμε να είμαστε σωστά ενημερωμένοι πριν από μία ψηφοφορία στην Ολομέλεια, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να θέσουμε και αυτό το στόχο της επικαιροποίηση ε, της μελέτης επιπτώσεων ή τουλάχιστον μια συμπλήρωση της μελέτης επιπτώσεων ανάλογα με τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε μια νομοθετική πρόταση. Αυτό είναι από οργανωτική άποψη ίσως το πιο δύσκολο σημείο για εφαρμογή, αλλά ο εξωτερικός έλεγχος, ε, η συμπερίληψη στο Συμβούλιο ε, Αξιολόγηση των Εκτιμήσεων και κάποιων ανεξάρτητων εταίρων, νομίζω ότι είναι εύλογες συστάσεις. Πάντως ε, ήταν καλό και το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρόλο φαίνεται ότι ασκούμε κριτική, Απλώς περιμένουμε κάποια βελτίωση και είμαστε λίγο πιο απαιτητικοί, αλλά δεν ε, απαξιώνουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ αυτά προς το παρόν και περιμένω τις συστάσεις. Ευχαριστώ. Ο σκιώδης συζητής, ο κύριος Μπέντζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή μας για το έργο του. Το σχέδιο γνωμοδότηση βρήθη θετικών σημείων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το γραφειοκρατικό άκθος και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λέμε ότι το διοικητικό άκθος της νέας νομοθεσία θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της μελέτη επιπτώσεων. Και μάλιστα η... θα πρέπει να γίνεται αντίστοιχη εφαρμογή και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι με κάποιες τροπολογίες μπορούμε να βελτιώσουμε τη γνωμοδότηση, γιατί ο, ο, ο αντίκτυπος α, ε, των συμφωνιών οικονομικές εταιρικής σχέσεις θα πρέπει να μελετηθεί δεόντως. Επίσης θα πρέπει να εξετάζονται οι επιπτώσεις συγκεκριμένων νομοθετικών ε, πρωτοβουλειών. Και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ε, να έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν τις προτάσεις τους πριν την οριστικοποίηση μιας μελέτης επιπτώσεων. Οπότε οι μελέτες επιπτώσεων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και μάλιστα εκτελεστικές ε, συνόψεις, ε, επιτομές θα πρέπει να είναι προσιτές. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από τους σοσιαλιστές η Σκιώδης, η συγχύτρια. Κυρία Μπαντία Ικουτσέτ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Τερέσα Ριέρα Μαδουρέλ, που βρίσκεται σε αποστολή. Θα, σα διαβάσω το κείμενό τη. Όπω είπα και στην προηγούμενη μου παρέμβαση, θα ήθελα να αναγνωρίσω την τεράστια προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελευταία πενταετία στα πλαίσια του Νομοθετή. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι απομένει σημαντικό περιθώριο λιγμών για την ενίσχυση τη διαδικασία των εκτιμήσεων, των επιπτώσεων. Η ομάδα μου πιστεύει ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την παρούσα δομή της Επιτροπής Εκτίμηση Επιπτώσεων, γιατί η ανεξαρτητοποίηση ουσιαστικά κατακαιρματίζει το δικαίωμα πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι θεμέλιο λήθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, λέμε να συμπεριλάβουμε ένα τμήμα, ένα ποσοστό ανεξάρτητων εμπειρογνωμών στην Επιτροπή μελέτη επιπτώσεων, προκειμένου να βελτιώσουμε τη διαφάνεια και την ποιότητα τη όλη διαδικασία. Και αυτό θα προτείνουμε, συμπερίληψη ενό ποσοστού ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Επίση, θα πρέπει να εξετάσουμε τι εκτιμήσει επιπτώσεων ω μια ε, ζωντανή διαδικασία που θα πρέπει να επηρεάζει την νομοθετική διαδικασία από τη σύλληψη μέχρι την εφαρμογή τη. Γι' αυτό και η ομάδα μου θεωρεί σημαντικό να δημοσιεύονται και να τυχάνουν διαβούλευση και τα σχέδια μελετών επιπτώσεων πριν να οριστικοποιηθούν. Επίσης, είναι σημαντική μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα εξετάζει ε, τις οικονομικές συνέπειες και ιδιαίτερα τον αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα λαμβάνει υπόψη υγειονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε σε μια αμυγός οικονομική προσέγγιση των μελετών επιπτώσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μετσάρος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει διαφανής, χρειαζόμαστε τις ε, μελετές επιπτώσεων, οι οποίες θα λάβανε υπο, υπόψη πτυχές υπερβραδικές, πολιτικές και το καθεξής. Τον Νοέμβριο του 2006 δημιουργήθηκε αυτή η Επιτροπή για την μελέτη επιπτώσεων και σκοπός ήταν να βελτιωθεί η ποιότητα των μελετών επιπτώσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασφαλώς ε, στηρίζει τον στόχο αυτό. Θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των μελετών αυτών, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι σημαντικό να μειωθεί και το διοικητικό κόστος, το διοικητικό φόρτος. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι μελέτες αυτές επιπτώσεων θα περνούν από τακτικούς ελέγχους, προκειμένου να επηρεάσουν πραγματικά το πολιτικό γίγνεσθε, γιατί πολύ συχνά δεν διεξάγονται μελέτες επιπτώσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, κάνει ό,τι μπορεί για να διεξάγονται οι κατάλληλες μελέτες επιπτώσεων στις κατοχώρες, στη Σουηδία, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία. Οι μελέτες αυτές δεν διεξάγονται από τα Υπουργεία, από την κυβέρνηση, αλλά από εξωτερικές υπηρεσίες. Είναι σημαντικό αυτό και είναι σημαντικό οι μελέτες αυτές να θεωρούνται ως υποστήριγμα, όχι ως αντικατάστατο των αποφάσεων και είναι σημαντικό τελικά να συνδράμουν σε μια καλύτερη νομοθεσία. Και θα πρέπει να φροντίσουμε η Επιτροπή αυτή να δρά ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να διορίζονται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να διασφαλίζουμε ότι τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν λόγο και κατά τον ορισμό των ε, προϋπολογισμών των κονδυλίων. Και τέτοιες μελέτες χρειάζονται σε κάθε νομοθετική διαδικασία, ιδιαίτερα σε αυτές πολιτικής φύσεως. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Τούρμες, λέει ο Πρόεδρος. Thank you. Ευχαριστώ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι υπάρχει εκπρόσωπο εδώ στην αίθουσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί θα με ενδιαφέραν τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την πρότασή μας. Γιατί όλα αυτά που προτείνουμε τι επιπτώσεις, ε, τι θα έχουν ε, στις καθυστερήσεις. Γιατί για την οικονομική κρίση θα χρειαστεί ένα-δύο χρόνια να συντάξουμε τις μελέτες επιπτώσεων πριν περάσουμε στη δράση. Οπότε όλες αυτές οι προτάσεις ε, που καταθέτουμε θα πρέπει να είναι και εφικτές. Γιατί είμαι βέβαιος ότι μετά από 25 χρόνια εφαρμογής πολιτικής ε, του αόρατου χεριού, όταν έχουμε και σπάνι ε, πόρων, θα περάσουμε σε μια εποχή που θα χρειαζόμαστε περισσότερη νομοθεσία, φυσικά ευφύ νομοθεσία, έξυπνη νομοθεσία. Δεν συμφωνώ λοιπόν ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από τη διακυβέρνηση, ότι είναι περίτη ανάγκη. Φυσικά και έχουμε και κάποιους ε, ανθρώπους όπως τον Τζάιλς που προτιμούν λιγότερη Ευρώπη, θεωρούν ότι λιγότερη Ευρώπη είναι καλύτερη. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η προσέγγιση ούτε και στο παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας. Οπότε, αν θέλουμε μελέτες επιπτώσεων, θα πρέπει σίγουρα να βελτιώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος των οικονομικών πράξεων, αλλά η νομοθεσία δεν θα πρέπει να είναι μόνο φιλική προς επιχειρήσεις, θα πρέπει να είναι φιλική και προς τους πολίτες. Όχι μόνο τους πολίτες ε, αυτής της γενιάς, αλλά και των επερχόμενων γενεών. Συμφωνώ με την ε, ιδέα των σοσιαλιστών που λένε ότι όλες οι μελέτες επιπτώσεων θα πρέπει να μην έχουν μόνο οικονομική διάσταση οι μελέτε επιπτώσεων, αλλά και κοινωνική διάσταση. Και κάτι που ξεχνούμε πολύ συχνά στη χάραξη πολιτικών είναι ότι αμελούμε τι επερχόμενε γενιές, γιατί εμεί, ε, ω πολιτικοί σκεφτόμαστε κοντόφθαλμα, σκεφτόμαστε μόνο υπό το πρίσμα των επόμενων εκλογών, προσπαθώντα να βολέψουμε κάποια λόμπι, κάποια στρώματα του πληθυσμού ή κάποιε ομάδε πολιτών που μα είναι σημαντικέ ε, για τι επόμενε εκλογέ. Αλλά α μην ξεχνούμε και τις επόμενε γενιές τους απογόνους μας και να δούμε τι σημαίνει μία νομοθεσία ή παράληψη μίας νομοθετικής δράσης για τις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ, αλλά νομίζω, Κλοντ, ότι το θέμα τώρα δεν είναι αν θέλουμε πιο πολύ ή πιο λίγη η Ευρώπη, αλλά όταν ε, κατατίζουμε νομοθεσία να είναι καλύτερη νομοθεσία. Αυτό είναι το θέμα και έχει γίνει έντονη συζήτηση για τις επιπτώσεις ε, κατά πόσον τις γνωρίζαμε και τις ε, αντιλαμβανόμασταν πλήρως τις επιπτώσεις. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει βασική διαφορά μεταξύ ε, επιχειρήσεων και πολιτών. Και οι επιχειρήσεις, οι πολίτες είναι. Ο Τσάλ ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα. Η Επιτροπή. Υπάρχει κανείς ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ που θα μπορούσε να απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν. Ναι, έχουμε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όχι τους ειδικού για το θέμα αυτό άρα δεν μας εξυπηρετεί. Να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους της ε, Επιτροπής που βρίσκονται εδώ, αλλά να δώσουμε το λόγο στον Τζάιλς. Μπορώ μόνο να πιθανολογήσω ότι Αποουσιάζεται ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί βρίσκεται κάπου προσπαθεί να εκτιμήσει, να αξιολογήσει τι επιπτώσει τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτού του θέματο. Είναι κάπου και προσπαθεί να εκτιμήσει τι επιπτώσει ε, αυτή τη ε, ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστώ για τα επικοδομητικά σας σχόλια και περιμένω και τροπολογίες που θα τα αποτυπώνουν. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σχόλια. Το πρώτο ήταν της κυρίας Ριέρα Μαντουρέλ. Εγώ δεν μιλώ για μια ριζοσπαστική αλλαγή, για μια ρηξικέλευθη μετάβαση σε μια νέα διαδικασία και κατάργηση προηγούμενη. Όχι, αυτό θα ήταν επικίνδυνο. Απλώ προτείνω αλλαγή ορισμένων στοιχείων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή μια ανεξάρτητη σκέψη σε αυτή τη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να συμπλέψουμε τελικά ως προς το ποσοστό ανεξαρτησίας που θα θέλαμε να προσθέσουμε στην όλη διαδικασία. Το σχόλιο του αξιότιμου συναδέλφου Κλοντ Τέρμες είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ακούσαμε και την προηγούμενη φορά, αλλά διευρύνουν υπερβολικά τη συζήτηση από το τεχνικό ε, επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σε ένα πιο μεταφυσικό και πιο λυρικό. Μη φαντάζεστε ότι οι πολίτες διεκδικούν περισσότερη νομοθετική παρέμβαση, περισσότερη και μερική νομοθεσία, αλλά αυτό που περιμένουν οι πολίτες από εμά είναι να ελέγξουμε τις νομοθετικές διατάξεις για να δούμε ποιες είναι καλές και ποιες είναι εφαρμόσιμες και εφικτές. Ναι, άκουσα το σχόλιο. Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε αμυγός σε οικονομικέ πτυχέ, γιατί σίγουρα η νομοθεσία δεν έχει μόνο οικονομικό χαρακτήρα. Αλλά και το θέμα το οικονομικό είναι σημαντικό και η χρηματοδότηση είναι σημαντική. Όταν εξετάζουμε τις νομοθετικέ προτάσεις, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις οικονομικές τους συνέπειες. Και αυτό είναι σημαντικό Πάντως, πιστεύω ότι η πρόταση του Κλοντ για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή της γνωμοδότησης είναι μάλλον εκτός θέματος και δεν νομίζω θα επέλθει συντέλεια του κόσμου Κλοντ αν δεχτούμε την γνωμοδότηση έτσι όπως έχει. Αυτά και ευχαριστώ. Περιμένω τροπολογίες. Ευχαριστώ και κλείνω το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Να περάσουμε στο σημείο 11 τώρα πράσινη βίβλος για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λένα Έκιν, η συντάκτρια της γνωμοδότησης και της δίνω κατευθείαν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. this is, uh... Πρόκειται για μια πράσινη βίβλο. Ως εκ τούτου, καλό είναι να συζητήσουμε το μέλλον των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τα δάση είναι πολύ σημαντική αξία και οικονομική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν κοινωνική ιστορική διάσταση, αλλά έχουν και αξία αναψυχής, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι αναψυχής ή επιτρέπουν στον κόσμο να περάσει ευχάριστα ένα τίμα του ελεύθερου του χρόνου. Αν εξετάσουμε το ΕΠ στην Ευρώπη, η δασική βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 10%, άρα είναι σημαντική συμμετοχή των δασών και 9% της μεταποίησης ε, και του εργατικού δυναμικού καλύπτονται, απασχολούνται στην, στον δασικό κλάδο. Υπάρχουν, υπάρχει μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας γύρω από τα δάση και το, το δασικό κλάδο. Εκτελήσετε συζήτηση για το κατά πόσο διαχειριζόμαστε με λάθος τρόπο τα δάση. Αυξάνονται οι δασικές εκτάσεις. Στην Ευρώπη, ναι, 1% το χρόνο. Και μάλιστα την τελευταία πεντακονταετία. Στις σκανδιναβικές χώρες τέτοια ανάπτυξη παρατηρείται εδώ και 100 χρόνια. Ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, όσο μεγαλώνουν τα δάση, καταφέρουμε και να έχουμε ένα βιώσιμο κλάδο που γενικώ παγκοσμίω θεωρείται επίτευγμα. Γιατί τέτοια ανάπτυξη και άθηση των δασών μόνο στην Ευρώπη βλέπουμε. Ταυτόχρονα, αν δούμε το θέμα υπό το πρίσμα της βιώσιμης δασικής διαχείρισης και της προστασίας, βλέπουμε ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια βιοπικιλότητα των δασών και μια προσαρμοστικότητά τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών γιατί σίγουρα η θέρμανση του πλανήτη επηρεάζει και τα δάση. Και αυτό το παρατηρούμε και για ορισμένα είδη που αρχίζουν και μεταναστεύουν ε, προς βορρά. Στην πατρίδα μου αρχίζουμε και παρατηρούμε ένα είδος ε, σημίδας για παράδειγμα που πρώτη φορά εμφανίζεται τα τελευταία 100 χρόνια ή το βλέπουμε και σε έντομα που αρχίζουν και μεταναστεύουν προς βορράν όλο και περισσότερο. Για παράδειγμα, σκαθάρι της, των πεύκων ε, παρατηρείται σε περιοχές που δεν υπήρχε προηγουμένως. Και το θέμα των δασικών πυρκαγιών είναι τεράστιο και ακαθόδες φλέγων για χώρες του Νότου κυρίως. Δυστυχώς οι πυρκαγιές έχουν πλήξει τον Νότο και έχουν αναχθεί πλέον σε κοινωνικό πρόβλημα. Η πράσινη αυτή βίβλος δεν επιχειρεί τόσο προστασία, αλλά προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή. Φυσικά η προσαρμογή περιλαμβάνει και την προστασία, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα διάφορα είδη, τη χλωρίδα και την πανίδα και πώς συγκεντρώνουμε σημαντικές για μας πληροφορίες. Χρειαζόμαστε μια πραγματική στρατηγική των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και χρειαζόμαστε προδιαγραφές, στατιστικά στοιχεία, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε αρκετές γνώσεις για να αποτιμήσουμε την κατάσταση και να ξέρουμε τι γίνεται. Ο πρώτος πυλώνας της Πράσινης Βίβλου είναι η συγκέντρωση της γνώσης ε, των προδιαγραφών και των στατιστικών. Επικροτώ αυτή την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι πρόβλημα και σε διεθνέ επίπεδο. Ετοιμαζόμαστε τώρα για τις ε, διαπραγματεύσει ε, περί κλίματος που θα γίνουν στο Μεξικό το Δεκέμβριο. Και μάλιστα η διαχείριση των δασών αποτελεί προτεραιότητα της ε, ημερήσια διάταξης αυτής της συνδιάσκεψης. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί αποφάσεις για το περιβάλλον έχουν επιρροή και στη διαχείριση των δασών. Θα πρέπει λοιπόν να προετοιμαστούμε για αυτές τις συζητήσεις ε, και στον ΟΗΕ. Το πρόβλημα είναι ότι ορισμένα θέματα αποφασίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά στον τομέα αυτό ισχύει κυρίως η επικουρικότητα. Εγώ δεν είμαι κατά της επικουρικότητας, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα σε θέματα επιμόρφωσης, ε, ανταλλαγής γνώσεων, αξιοποίησης των βέλτιστων πρακτικών και φυσικά έρευνας. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε μία βιομηχανική πλατφόρμα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο με θέμα τα δάση, τη δασοκομεία. Θα πρέπει να παραμείνει γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα των δασών στις στην ενδιάμεση αναθεώρηση για το πρόγραμμα, 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά εν ώψη και των διαπραγματεύσεων για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Σε, πολλούς τομείς, σε, πολλούς, σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, τα δάση είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αποτελούν και βάση για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας και δικαιωμάτων κυριότητα των δασών, γιατί και τα δικαιώματα κυριότητα είναι πολύ σημαντικά. Η διαχείριση των δασών στην Ευρώπη γίνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο. Κάθε χώρα έχει υιοθετήσει έναν ιδιόμορφο τρόπο για τη διαχείριση των δασών και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων για τα δάση. Και αν δείτε το ιστορικό της ε, νομοθεσίας περί δασών, βλέπετε ότι έχουν γίνει πολλά σφάλματα, αλλά ταυτόχρονα έχουν εφαρμοστεί και πολύ καλές πρακτικές στην Ευρώπη. Στην έκθεση αυτή λοιπόν προσπαθώ να προσεγγίσω το θέμα υπό ένα βιομηχανικό πρίσμα. Παρακολούθησα και την χθεσινή συζήτηση στην Επιτροπή της Γεωργίας. Φυσικά είχε διαφορετικό περιεχόμενο από τη δική μας. Και μάλιστα είμαι και σκιώδη συγγήτρια της έκθεσης ε, στην Επιτροπή Γεωργίας και θα προσπαθήσω να καταφέρω τη συμπερίληψη κάποιων τμήματων της γνωμοδότησής μου και στην τελική έκθεση του εισηγητού της Επιτροπής Γεωργίας. Όταν ασχολείται κανείς με τα δάση, διαπιστώνει ότι ελάχιστοι είναι οι υπάλληλοι της Επιτροπής που έχουν ε, βαθιά γνώση για τα δάση. Ελάχιστοι εμπειρογνώμονες για τα δάση υπάρχουν στις διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν ξέρω πώς θα καλύψει αυτό το κενό στα, στη στελέχωσή της στις διάφορες γενικές διευθύνσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πρόεδρε και μακάρι να εκδηλωθεί όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για θέματα δασών. Ευχαριστώ πολύ και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα συμβεί. Να πω ενημερωτικά κάτι για το προηγούμενο σημείο που ξέχασα. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για την έκθεση του Giles είναι η 5η Οκτωβρίου. Είναι σαφές μεν, αλλά οφείλω να το αναφέρω. 5η Οκτωβρίου προθεσμία. Λένα. Ναι. Αν θα μπορούσε η Γραμματεία να ενημερώσει τα μέλη για το χρονοδιάγραμμα, των άλλων επιτροπών. Για τη δική μου έκθεση μιλώ. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, να περάσουμε τώρα στη συζήτηση για την έκθεση για τα δάση. Η Ο σκιώδης συζητητής ε, Πάνταρ. Ευχαριστώ. Ε, καλωσορίζω το κείμενο και συμφωνώ με τα περισσότερα σημεία ως εισηγητή των σοσιαλιστών έχω και εγώ κάποια σχόλια να κάνω. Καταρχάς για το σημείο 1 σε ό,τι αφορά την διατήρηση και τη βελτίωση των λειτουργιών των δατσών. Πέρα από την βιοπικιλότητα θα υπάρξει σημασία και θα δοθεί προσοχή και σε άλλες πτυχές των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται έντονη συζήτηση ε, για τις οικολογικές υπηρεσίες. Κατά δεύτερον, η Ευρώπη θα πρέπει να καταρτήσει πρωτοβουλίες σε όλο το φάσμα της Ευρώπης. Για το σημείο 4 τώρα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι <laughs> χρειάζεται μια δίκαιη κατανομή του συστήματος RED. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει χωρίς μεταρρύθμιση του κλάδου και της διαχείρισης του κλάδου. Και επίσης προτείνω κάποιες τροπολογίες για την βιώσιμη διαχείριση των δασών, γιατί υπάρχουν διαφορές ό,τι αφορά την εφαρμογή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα τούτο, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις συζητήσεις που διεξάγονται μέχρι το 2013 για την διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τα μέτρα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε μια σωστή διαχείριση των δασών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμπερτς είναι επόμενος ε, ειδικός, ειδικός, ειδήμονας. Τώρα μην υπερβάλλουμε κιόλα, λέει ο κύριος Λάμπερτ να συνεχίσω και να υποστηρίξω αυτά που είπε ο συνάδελφος για την πτυχή της βιοπικιλότητας, γιατί βρισκόμαστε στο έτος της βιοπικιλότητας, αλλά μιλάμε για θέμα προσαρμογής. Κοιτώντας την βιοπικιλότητα των δασών είναι η πιο ευάλωτη, είτε στα ακραία καιρικά φαινόμενα, και αυτό το είδαμε και στη Γαλλία, στο Βέλγιο, σε όλες τις χώρες, όπου μεγάλες θύελες ήρθαν από πλευράς Ατλαντικού και ουσιαστικά εξάλληψαν ε, είδη ζώων, είτε από επιθέσεις εντόμων. Αν δεν υπάρχει βιοπικιλότητα, τα δάση δεν μπορούν να τα επεξέλθουν. Άρα θα πρέπει να τονιστεί το σημείο αυτό και είμαστε ε, Επιτροπή Βιομηχανίας. Άρα θα πρέπει να τονίσουμε την πτυχή της ε, προστασίας των πόρων και της οικονομικής αξίας. Γιατί γνωρίζουμε ότι τα δάση, α, αν τα δάση καταστραφούν από θύελε και από μάστιγες, αυτό θα έχει και οικονομικό αντικτύπο. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερον, να δούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν Έχουμε την τάση να καταρτίζουμε νέες πρωτοβουλίες χωρίς απαραίτητα πάντα να εξετάζουμε τον αντίκτυπο των ε, τρέχουσων ε, πρωτοβουλειών. Θα πρέπει να κοιτάξουμε το σχέδιο δράσης για την δασοκομεία και άλλες σχετικές ε, νομοθεσίες, την στρατηγική για την δασική διαχείριση που έχει εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε κατά πόσον έχει πετύχει κάτι, έχουν πετύχει κάτι αυτές οι πολιτικές. Να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια ανασκόπηση προκειμένου να βελτιώσει τον αντίκτυπο της ισχύουσας νομοθεσίας. Αυτά είναι τα δύο σημεία που ήθελα να τονίσω. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε με όσα μας είπε η Λένα. Δεν έχουμε σημεία διαφωνίας, απλά θα θέλαμε να προσθεθούν κάποια σημεία επιπλέον. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. πολύ οξυδερκής οι παρατηρήσεις και αξιόλογη γνωμοδότηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγητρία που αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των δασών στην Ευρώπη και τη σημασία της πράσινης βίβλου. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω, να επαναλάβω αυτό που μας είπε για τα δάση που καλύπτουν 42% της συνολικής επιφάνειας. Δεν μπορούμε να υποτιμούμε λοιπόν την σημασία τους να πω δύο λόγια για το περιεχόμενο της πράσινης βίβλου και ποια θα θέλαμε να είναι τα αποτελέσματά της. Η νέα στρατηγική των δασών ε, συνοδεύεται και από ένα σχέδιο δράσης για τα δάση. Και οι βασικές δράσεις για το νέο σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δάση περιλαμβάνει διάφορα μέτρα προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επίσης, αναγνωρίζουμε την ανάγκη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού, πανευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης των δασών και ανάγκη της προστασίας φυσικά των ευρωπαϊκών δασών. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει μια λευκή βίβλο προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές και εκεί επισημάναμε την ανάγκη να ασχοληθούμε με την προστασία των δασών υπό το φως, υπό το πρίσμα των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών που ήδη γίνονται αισθητές σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Η Πράσινη Βίβλος παρουσιάζει την κατάσταση των ευρωπαϊκών δασών, τη λειτουργία τους, τον αντίκτυπο των κλιματικών αλλαγών στα δάση, όπως έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής και κάποιες προβλέψεις. Ε, αναλύουμε τους ισχύοντες μηχανισμούς για την προστασία των δασών, καθώς και τις πηγές πληροφόρησης που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και επίσης ε, ξεκινάει μια συζήτηση για τα θέματα αυτά. Είμαστε παρκώς προετοιμασμένοι για τις κλιματικές αλλαγές και όχι μόνο για τις κλιματικές αλλαγές αλλά και τις επιπτώσεις τους ε, και το πώς ε, επηρεάζουν αυτές τα δάση. Είναι επαρκείς οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Τι μπορεί ε, να προσθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους ισχύοντες μηχανισμούς. Υπάρχει λόγος και χώρος για μια επιπλέον δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα αυτό. Ξεκίνησε μια διαβούλευση με πλούσια συμμετοχή. Λάβαμε 261 προτάσεις από διάφορους ενδιαφερόμενους εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε την επεξεργασία όλων αυτών των συνεισφορών, οπότε δεν έχουμε καταλήξει συμπεράσματα αυτής της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε. Τώρα εκτελήσεται αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης των συνεισφορών και έχουμε λάβει και τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Από τη στιγμή που θα επεξεργαστούμε και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μασενκίβιτς, τον οποίο ξέχασα προηγουμένως. Ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη χαρά ε, λαμβάνω τη γραμματότητα της κυρίας ΣΕΚ και τα έγραφα γενικώ ε, για την έναρξη συζήτηση περί προστασίας των δασών και της κατάστασης ε, των ε, δασών. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για την δασική οικονομία. Αναβαθμίζεται έτσι η κατάσταση των δασών και της δασοκομείας, γιατί είναι σημαντικό κοινωνικό ζήτημα η προστασία των δασών. Τα δάση έχουν πολλούς, πολλούς ρόλους για παράδειγμα, απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε η προστασία τους ε, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, βιωσιμότητά τους, αλλά να περισσώσουμε και τη βιοπικιλότητα ε, των δασών. Γιατί 70% αυτής της βιοπικιλότητας λαμβάνει χώρα στα δάση. Γι' αυτό θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε με ορθολογικό τρόπο, γιατί τα δάση σχετίζονται και με πολιτιστικές αξίες, με οικονομικές, κοινωνικές, αλλά και με θέματα απασχόληση. Είναι πολυλειτουργικά τα δάση. Το θέμα του, της του περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με τα δάση. Τα δάση δεν έχουν μόνο αξία για την υλοτομία τους, αλλά έχουν πολύ επίπεδη αξία. Επίσης είναι σημαντικά για την ίδια την κοινωνία. Η δασική οικονομία και μια σωστή δασική οικονομία δεν ε, εξασφαλίζει μόνο ε, την ε, αποφυγή των θεομηνιών ή των πλημμυρών, αλλά εξασφαλίζει και ένα καλύτερο περιβάλλον. Περιμένουμε τη συνέχεια της συζήτησης ε, με διάφορους ενδιαφερόμενους γιατί θα πρέπει να προβούμε σε μια εξισορρόπηση μεταξύ των ε, δικαιωμάτων προστασίας και των δικαιωμάτων κυριότητας γιατί υπάρχουν διαφορετικά συστήματα. Κάθε χώρα έχει διαφορετικά ε, είδη δασών. Μερικές φορές τα δάση είναι παλιά δάση ε, και όσο πιο παλιά είναι τα δάση, τόσο λιγότερη δυνατότητα έχουν απορρόφησης διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην αναδάσωση. Επίσης, από πρακτική άποψη, θα πρέπει να καθορίσουμε κάποιες ε, ε, αρχές για να βελτιώσουμε την απορρόφηση από τα δάση του διοξιδίου του άνθρακα. Συμφωνώ με την ε, κυρία εισηγήτρια ότι η αρμοδιότητα για την ε, δασική οικονομία θα πρέπει να παραμείνει στα πλαίσια της επικουρικότητας στα χέρια των ε, ευρωπαϊκών χωρών. Βέβαια, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στο συντονισμό. Θα πρέπει να στηρίξουμε τη διαδικασία προσαρμογής των δασών στις κλιματικές αλλαγές. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να βοηθήσουμε τα δάση ε, θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες ε, και με οικονομικούς τρόπους για να προσαρμόσουν τα δάση τους στις κλιματικές αλλαγές. Επίσης θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιους κοινούς μηχανισμούς για τα δάση, όχι μόνο για να στηρίξουμε την πολυεπίπεδη δασική οικονομία, αλλά να βρούμε κάποιους τρόπους ε, για να στηρίξουμε την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα λοιπόν να σας προσκαλέσω και στην έκθεση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα που αφορά τα δάση και την προστασία της φύσης, του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και να δώσω το λόγο στη συνάδελφο ΕΚ για να κλείσει. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τα πολύ χρήσιμα σχόλια που κάναν. Είμαι βέβαιη ότι θα είναι πολύ καλή η συνεργασία μας επί του κειμένου. Κάποια σχόλια επιτρέψτε μου για τις παρατηρήσεις που κάνετε. Φυσικά η προσαρμογή και η βιοπικιλότητα αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία και χρειάζονται, χρειάζονται και τα δύο. Πριν από κάποια χρόνια επισκέφθηκα τον Καναδά και πέταξα με αεροπλάνο πάνω από τις τεράστιες εκτάσεις πάνω από το όρος καθάριτων πευκών που είχε καταστραφεί. Ήταν πραγματικά φρικτό. Εκατοντά τετραγωνικά χιλιόμετρα είχαν καταστραφεί. Αν αυτό συμβεί και σε εμά, μπορούμε να ξεχάσουμε οποιαδήποτε διαχείριση των δασών. Πρόκειται για μια σοβαρή απειλή και για τις TLS. Μένω στα προάστια μιας περιοχής που πλήχθηκε πάρα πολύ άσχημα πριν από κάποια χρόνια. Και βλέποντας τον αντίκτυπο τέτοιας, τέτοιων καταστροφών, συμφωνώ ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά. Το θέμα είναι πώς θα το συνδυάσουμε με θέματα διοκτησίας και εμ, επικουρικότητας. Θεωρώ ότι χρειάζεται πληροφορίες, γνώση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει αυτή η γνώση να, να διατεθεί και στις κυβερνήσεις αλλά και σε αυτούς που διαχειρίζονται τα δάση. Αυτά είναι κάποια προβλήματα ενδεικτικά. Να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να με βοηθήσει στο εξή. Εξετάζοντα την νομοθεσία που ισχύει για την κοινή αγροτική πολιτική, πρέπει να πω ότι είναι αντιπαραγωγική. Δεν βοηθά τους στόχους που προσπαθούμε να πετύχουμε σε ό,τι αφορά την προστασία, την προσαρμογή και την επέκταση των δασών λόγω της αξίας που έχουν για την βιοπικιλότητα και για το κλίμα. Εδώ και χιλιάδες ε, χρόνια στη Σουηδία βοσκούν τα ζώα στις κοιλάδες και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται και λέει ότι αυτό δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Μιλάμε για εκτάσεις όπου μπορεί να υπάρχουν 80 δάση ανά ενώ η Επιτροπή προδιαγράφει 50 ανά εκτάριο. Δηλαδή τι κάνουν τώρα οι αγρότες στην Σουηδία, κόβουν τα δέντρα σε, παραδοσιακούς, ε, σε παραδοσιακές περιοχές, εξετάζοντας θέματα βιο Μιλάμε για περιοχές όπου υπάρχουν λουλούδια, χόρτα τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Και ουσιαστικά είναι αντιπαραγωγικός ο τρόπος εργασίας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πολιτικά. Θα αλλάξουμε τα ζητήματα δασικής διαχείρισης ή γεωργικής πολιτικής. Γιατί από πλευρά ευρωπαϊκού συστήματος πρέπει να πω ότι το σύστημα φαίνεται ανόητο. Θέλουμε να πετύχουμε δύο διαφορετικά πράγματα και είναι αδύνατο να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Είναι πρακτικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος, αν θέλετε, ένα γενικότερο υπόβαθρο ως προς τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε για τα θέματα αυτά. Επίσης από πλευράς ε, κλιματικής. Φυσικά, τα δάση αποτελούν πηγή εναλλακτικών ενεργειών. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε και την πτυχή αυτή και να καταλάβουμε ότι από πλευράς κλιματικής η προστασία των δασών Υπάρχει και η πτυχή της ε, σύψης των ε, ε, δασών, των δέντρων, του ξύλου, η οποία ε, εκλείει διεξίδιο του άνθρακα σε μεγάλα ποσοστά. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι έχουμε την μέγιστη την αντιπαραγωγή γιατί αυτό επηρεάζει την επιτευξή των κλιματικών στόχων και θα μπορούσαμε να έχουμε διαχείριση και στον υπόλοιπο κόσμο, και οι στόχοι που έχουμε θέσει στην ε, Βόρεια Ευρώπη από μόνοι του, σε ό,τι αφορά τα δάση, από μόνοι τους θα πετύχαιναν του στόχου που έχουμε θέσει για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και θα πρέπει να υπάρξει προστασία, προσαρμογή, αλλά και παραγωγή. Αυτή την ισορροπία προσπάθησα να πετύχω στην έκθεσή μου. Και πραγματικά ανυπομονώ να συζητήσω και με τους σκιώδεις συζητητές, γιατί θεωρώ ότι έχουμε κοινέ αξίες στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 12 Οκτωβρίου, 12 η ώρα είναι η εκταλεκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Για να ψηφίσουμε 8 και 9 Νοεμβρίου στην ε, Επιτροπή μας να δούμε και πότε θα γίνει και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντο και να δούμε πότε θα περάσει στην Ολομέλεια. Μάλιστα, λοιπόν, ολοκληρώθηκε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Να περιμένουμε πέντε λεπτά για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία ή να ξεκινήσουμε. Ή θέλετε μήπως να ξεκινήσουμε με την έκθεση Μπέντσεν. Αν δεν έχουν έρθει ακόμα οι σκιώδεις. Ε, εντάξει, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Πέντε λεπτάκια και μετά θα ξεκινήσουμε με τις πληροφορίε. Ladies και gentlemen, we can start. Έχετε σας την να ξεκινήσουμε. Αν έχουν έρθει όλοι οι συνάδελφοι, να, ξεκινήσουμε με την έκθεση Καρβάλιο πολύ μεγάλη έκθεση με πολλές τροπολογίες. Ευτυχώς, η συνάδελφος μας ε, διευκόλυνε λίγο στην εργασία μας. Και έχουμε και κάποιες ε, συμβαστικές προτάσεις να ψηφίσουμε. Να ξεκινήσουμε με το 5α. Μετροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Τρία Συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποφασιστική. Εγκρίνεται. Πρόεδρε, δεν είμαι βέβαιος, Πρόεδρε, ότι η Ρέτζι 2 καταπίπτει πλήρως, γιατί αναφέρεται καταπίπτει μόνο το πρώτο τμήμα, εάν εγκριθεί η συμβαστική 3. Πριν το 5, πριν την τροπολογία υπαριθμών 5, ναι, δίκιο έχετε, λέει ο Πρόεδρος. Αλλά μου λέει η γραμματεία ότι το υπόλοιπο τμήμα της τροπολογίας θα το κοιτάξουμε αργότερα σε άλλη τροπολογία. Πάμε λοιπόν στη συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 10. Και η, 40 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 36. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 38 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Με προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 53. Ακαλύπτεται. Η 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 56 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. 57. Ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 με προφορική τροπολογία. Την έχετε την προφορική τροπολογία μπροστά σα. Δεν υπάρχουν ερωτήσει. Με προφορική τροπολογία υπέρ λοιπόν. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμόν 9 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 70 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 72 υπέρ. Α, δεν είναι απαραίτητο. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 12. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 81 δεύτερο τμήμα γιατί το πρώτο αποσύρθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ με προφορική τροπολογία Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Απόχες. Να τα, το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για τη συμβαστική υπαριθμών 11. Ψηφίστε παρακαλώ.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 29 υπέρ, 20 κατά, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 93 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 96 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, αποσύρεται, 102 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι. Α, 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Κοντ 2 Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκα... 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115. Υπέρ κατά. Άποχες, απορρίπτεται. 116 υπέρ. Κατά. Άποχες, εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Άποχες, απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Άποχες, απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Άποχες, απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Άποχες, Απορρίπτεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Δεν είμαι σίγουρος για την 122. Παρακαλώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Board is closed. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται 123 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται 124 υπέρ. Α, συγγνώμη, πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, να το ελέγξουμε παρακαλώ για το δεύτερο τμήμα της 124 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. Ρέγγι. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας. <clears throat> Πέρασε και το αποτέλεσμα το βλέπετε. Εγκρίνεται με συντριπτική πλειοψηφία. Χαρτίρια στην εισηγήτρια και θα αποτελέσει σημαντική βάση για τι μελλοντικέ συνεργασίε. Η έκθεση αυτή, η επόμενη έκθεση του κυρίου Φράγκο, έχετε μπροστά σα δύο υπέρ. Κατά. Δύο παρακαλώ υπέρ. Κατά. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 5. Σε τμήματα τώρα στην 9. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπληκτή επόμενη, η 11, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, Δεύτερο τμήμα, λέει ο πρόεδρο. Α, συγγνώμη. Η 12, λέει ο πρόεδρο. Η 12, η 12, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην 1. Υπέρ. Α, όχι, λέει ο πρόεδρο. 12? 12 is adopted, so we do not ah, it sticks. I must vote on the original vote. No, no, we do not no, it's four. Ναι, καταπίπτει, λέει ο πρόεδρος. Τι γίνεται. Δίκιο είχα. Παρακαλώ, λίγη ησυχία. Η ένα, παρακαλώ. Υπέρ, κατά. Άποχες, απορρίπτεται. Η έξι, αποσύρθηκε. Επτά, υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 14. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. πίπτη 16. 17. Υπέρ. Κατά. Και πάλι να ψηφίσουμε πάλι 17 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Άποχες. Ε, εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 20 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται 22 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 καταπίπτει καταπίπτει 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 όχι English What was problems? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ρωτάει ο πρόεδρο. 24. Καταπίπτει 24. Διαφωνείτε. Να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 24 παρακαλώ. Ηλεκτρονικός ε, έλεγχο. Ένα ψηφοφορίας. Board is closed. And... Πέρας. Απορρίπτεται. Σαφές, σαφές. 25. Δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. 26. Υπέρ. Για την 26. Κατά. Ε, αποχές. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 κατά αποχές εγκρίνεται. 29, 29 καταπίπτει. 30 υπέρ κατά. Να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 30 ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας για την 30. πέρασε.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 και ποιο κέρδισε τελικά, λέει ο πρόεδρο. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρα. Είναι σαφέ λοιπόν το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 14, για την αναθεώρηση του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση και να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Μπέντσεν, τον εισηγητή. Και είναι και ο μοναδικός που θα πάρει το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να πω σε όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις συζητήσεις και την επεξεργασία αυτού του θέματος, ότι πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Χθες πάλι μιλήσαμε για την ενεργειακή μας στρατηγική μέχρι το 2020. Σήμερα Έχουμε την έκθεση για την αναθεώρηση του προγράμματος δράσης για την ενεργειακή απόδοση. Η Επιτροπή ετοιμάζει τις προτάσεις της και ελπίζω να ετοιμάσουμε μια έκθεση εμπεριστατωμένη ώστε το Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία να αποστείλει ένα ηχηρό μήνυμα προς την Επιτροπή. Πολλές οι απόψεις που εκφράστηκαν, πολλοί εδώ και οι συνομιλητές μας, αλλά ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια κοινή θέση απόλυτα συμμεριζόμενη από τους συναδέλφου. Ένα από τα ζητήματα είναι η συμμόρφωση και ένα άλλο η υλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας. Το ζήτημα είναι πού βρισκόμαστε σήμερα. Ποιους στόχους έχουμε ήδη επιτύχει, ποια είναι η νομοθεσία που βρισκομαστε σημερα Ποιου στοχους εχουμε ηδη επιτυχει υλοποιείται στα κράτη-μέλη και ούτω καθεξής. Οι μεγάλες προκλήσεις των υποδομών επίσης είναι ένα θέμα. Πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε ανανέωση των συστήματων όπως τα ευφυή δίκτυα, η ευφυής μέτρηση και η αποθήκευση ενέργειας που θα ε, διευκολύνουν και θα εξυπηρετήσουν την, απόδοση, την ενεργειακή απόδοση. Για τα κτίρια, τον τομέα τον κατασκευαστικό Ήδη έχουμε ένα σχετικό νόμο, όμω πρέπει να κάνουμε κάτι και για τα υπάρχοντα κτίρια. Το 40% τη ενέργεια καταναλώνεται από αυτά τα κτίρια. Επίση, για το IST και την ε, ενεργειακή ετικετοθεσία καθώ και τον ενεργειακό σχεδιασμό υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι η χρηματοδότηση. Έχουμε πολλέ δυνατότητε μεν, όμω η τραπεζική αγορά έχει παγώσει. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα κονδύλια και πολύ περισσότερα ποσά και επενδύσει σε αυτόν τον τομέα. Πάντω, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στι 4 Φεβρουαρίου θα συζητήσουν τα ενεργειακά ζητήματα και πρέπει να πω ότι η ενεργειακή απόδοση είναι ο φθηνότερος τρόπος για να περιορίσουμε και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πρέπει λοιπόν να περιορίσουμε την εξάρτησή μας από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Εδώ μιλάμε για ασφάλεια της παροχής και ενεργειακή απόδοση Υπάρχει λοιπόν μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Είμαι έτοιμος να καταγράψω τα σχόλιά σας και να συμμετάσχω σε όλες τις συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά σας και την εισαγωγή που κάναμε. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Τόμσον που είναι η σκιώδηση συγκεκριά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον ε, συνάδελφο Μπένσεν για το σχέδιο έκθεσή του. Η έκθεση συμπεριλαμβάνει πολλά σημαντικά στοιχεία για δράσεις προς αποτελεσματικότερη ενεργειακή απόδοση στην Ευρώπη. Ωστόσο, ήθελα να προσθέσω τέσσερα σημεία, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Η δεσμευτική στόχη, η ενεργειακή ένδυα, η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού και η χρηματοδότηση. Πρώτον, θα πρέπει να επιμείνουμε σε δεσμευτικούς υποχρεωτικούς στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας. Πιστεύω ότι ο στόχος του 20% μέχρι το 2020 είναι και ρεαλιστικός και φιλόδοξος. Ο δεσμευτικό χαρακτήρα των στόχων είναι καθοριστική σημασία, διότι θα είναι το πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενεργειακή Απόδοση. Χωρί τέτοιου στόχου δεσμευτικού, το πλαίσιο Τη ενεργειακή απόδοση και το πρόγραμμα δράση. θα είναι απλά λόγια και όχι πρόγραμμα δράση. Αυτό το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Επί χρόνια είχαμε στόχους που δεν ήταν δεσμευτικοί και δεν είχαμε αποτέλεσμα. Η ομάδα S&D θα υποβάλει μάλλον συγγνώμη, σοσιαλιστές θα υποβάλουν ε, τροπολογίες προκειμένου να βελτιωθεί η έκθεση. το Κοινοβούλιο είναι φιλόδοξο προς τους στόχου τους και θέλουν, θέλει να πιέσει την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικού στόχου ω το τέλο της χρονιάς. Έπειτα, έχω τονίσει επανειλημμένω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην ενεργειακή ένδυα ένα στοιχείο που δεν συμπεριλαμβάνεται στην, ε, στο σχέδιο έκθεση. Η ένδυα τη ενέργεια είναι ένα βασικό πρόβλημα για πολλά κράτη τη Ευρώπη, ιδίω τα νέα. Μια από τι μεγαλύτερε λοιπόν προκλήσει για το μέλλον είναι ότι η ενεργειακή ένδυα για τα καύσιμα θα επηρεάζει το εισόδημα των οικοκυριών, εφόσον μεγάλο μέρο του εισόδηματο αυτού θα δαπανάται για την ενέργεια. Πολλοί από του κατοίκου ε, στο πληρώνουν περισσότερο από 50% του εισοδήματό του για την ενέργεια. Η εμφάνιση λοιπόν της ενεργειακής ένδυας στην Ευρώπη είναι ένα σοβαρό φαινόμενο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να δούμε πώς θα την καταπολεμήσουμε αυτή την ένδυα και επίσης πρέπει να ζητήσουμε να αναλυφθεί δράση από την πλευρά του κοινού. Πρέπει να δοθούν κίνητρα προκειμένου να μειωθεί η δαπάνη ενέργειας Και επειδή για του φτωχότερου ιδίω τα κτίρια τα οποία διατίθενται, είναι αυτά που από την άποψη τη ενεργειακή απόδοση είναι τα λιγότερο αποτελεσματικά. Και η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ενεργειακή απόδοση. Πρέπει να ε, επικεντρωθούμε στι δεξιοτεχνίε και τι δεξιότητε και την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, την γνώση των νέων τεχνολογιών, την ε, εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά για τι φιλοδοξίε μα για την εξοικονόμηση ενέργεια. Πρέπει να κάνουμε σοβαρέ επενδύσει και στου ανθρώπου, όπω και στι τεχνολογίε. Τέλος, Θέλω να επικεντρωθώ στην χρηματοδότηση. Είναι θετικό ότι το σχέδιο έκθεσης αναφέρει διαφορετικού είδους μέτρα που θα μπορούσαν να αναλυθούν για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης. Το θέμα είναι όμως πώς μπορούμε να έχουμε κίνητρα για να βελτιώσουμε την ενεργειακή συμπεριφορά των πολιτών. Ε, το πρόγραμμα ΕΣΚΟΣ και παρόμοια προγράμματα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω. Θα ολοκληρώσω εδώ, αλλά ε, με τα χαρά να έχω περαιτέρω διαπραγματεύσει με τον εισηγητή και του υπόλοιπου συναδέλφου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Πέρα από αυτά που μας είπε και η σκιώδη εισηγήτρια, θα ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία φυσικά σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ενδία, αλλά και να συνδεθεί αυτό και με την ε, συνολική τιμή της ενέργειας και φυσικά αυτό συνδέεται και με την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα πρέπει να συνδεθεί αυτό και με την ε, μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αλλά οι τιμές ε, και την ενέργεια έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σημαντικά. Σε κάποιες χώρες περισσότερο από τις άλλες. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολεί. Αυτό θα πρέπει να συνδέσουμε. Και αυτό τι σημαίνει επίση ότι το ευρύ κοινό θα υποστηρίξει τέτοια μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και κατά δεύτερον μέσα στην έκθεση μιλάμε για έξυπνε λύσει. λύσεις ICT για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε ε, τα θέματα ενεργειακής ένδυας. Πολύ είναι καλό αυτό το smart meeting, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα μέτρα πολλές φορές ε, αυξάνουν το κόστος της ενέργειας, δυστυχώς. Να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Και τέλος, να τονίσουμε τα μέτρα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας και σε ό,τι αφορά φυσικά τα αριθμητικά ταμεία και τα λοιπά ταμεία και φυσικά η έκθεση επί της οποίας ε, εργαζόμαστε. Ελπίζουμε να περάσει σε πρώτη ανάγνωση. Ελπίζουμε όλα αυτά τα μέτρα να συμβάλλουν προκειμένου να είναι πιο διαφανής η αντιμετώπιση της, του θέματος. Και τέλος, μιλάμε με νέους και ατομικούς τρόπους για συστήματα τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων σχεδίων για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτά και θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω τον εισηγητή και θεωρώ ότι θα συμβάλλει σημαντικά η έκθεση αυτή προ τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εισηγήτρια. Um, Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπένσεν για την συνεργασία του πραγματικά διευκόλυνε του σκιώδει εισηγητές και μπορέσαμε να έχουμε διεξοδική συζήτηση του θέματο. Σα ευχαριστούμε λοιπόν. Συμφωνώ κατά πολύ με τον κύριο Μπένσεν ότι πρέπει να έχουμε μια έκθεση ισχυρή και περιστατωμένη, διότι όλοι νομίζω συμφωνούμε τελικά. Πρέπει να πω βέβαια ότι απογοητεύτηκα όταν είδα το πραγματικό κείμενο του σχεδίου έκθεση, το τελικό κείμενο, διότι είναι κάπως ήπιο το τι ζητά και απαιτεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Την τελευταία φορά το Κοινοβούλιο πραγματικά επηρέασε το πρόγραμμα δράση ενεργειακή απόδοση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι η Επιτροπή αναγκάστηκε να κάνει πράγματα που αρχικά δεν τα προέβλεπε, όμως ενθαρρύνθηκε να τα κάνει ε, χάρη στην ε, ενεργό δράση του Κοινοβουλίου. Αυτό που να ξαναγίνει λοιπόν τώρα. Και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη και το χρονοδιάγραμμα για την έκθεσή μα, τη στιγμή που ετοιμάζεται. Έχουμε ήδη μηνύματα από την Επιτροπή. Δεν έχουμε μάλλον επαρκή μηνύματα από την Επιτροπή για το πότε θα είναι έτοιμο το πρόγραμμά του. Είναι λοιπόν κέρια σημασία να παραμείνουμε στο αρχικό μα χρονοδιάγραμμα, γενικότερα για το πρόγραμμα δράση, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χάσουμε αυτή την ευκαιρία να ασκήσουμε πίεση όταν μπορούμε να επηρεάσουμε πραγματικά το τι θα, πώς θα διαμορφωθεί το περιεχόμενο του προγράμματος της Επιτροπής. Τώρα κάποιους τομείς στους οποίους θα ήθελα να ενισχυθεί η έκθεση. Σε ένα-δυο σημεία νομίζω ότι είναι λίγο εκ, ε, εκτός ε, επικαιρότητα. Και σε ό,τι αφορά την ε, υλοποίηση, νομίζω η έκθεση δεν δίνει υπαρκή έμφαση στο πώς θα πρέπει να παρακολουθούμε την Επιτροπή για το τι ε, έργο έχει γίνει ήδη στο παρελθόν για τα προγράμματα χρήσης της ενέργειας. Υπάρχει ένα πραγματικό χρονοδιάγραμμα που έχει υλοποιηθεί με μεγάλο κόπο και αυτή τη στιγμή δεν παρακολουθείται στενά. Παρομοίως λοιπόν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνονται από την Επιτροπή και η Επιτροπή θα πρέπει συνεχώς να προτείνει βελτιώσεις στα εθνικά προγράμματα ενεργειακής χρήσης και απόδοσης. Αυτό πήγε καλά με τα προγράμματα δράση για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, όμω πρέπει να πιέσουμε την Επιτροπή να κάνει τι ίδιε βελτιώσει ε, και να χρησιμοποιήσει αυτά τα διδάγματα και στο πρόγραμμα, στα προγράμματα δράση ενεργειακή απόδοση. Για του δεσμευτικού στόχου, ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικέ ε, απόψει ε, στο Κοινοβούλιο για το τι είδου δεσμευτικοί στόχοι είναι απαραίτητοι. Πάντω, σίγουρα κάτι τέτοιο χρειάζεται, διότι η Επιτροπή, ο Επιτρόπο μάλλον, έχει δείξει και έχει εκφράσει ότι, την άποψη ότι χρειάζονται δεσμευτικοί στόχοι για τον τομέα των κτηρίων. Δεν πρέπει λοιπόν εμεί εδώ να φανούμε ε, επιφυλακτικοί και λιγότερο φιλόδοξοι την ίδια την Επιτροπή. Ιδιαίτερω θα πρέπει κάτι να κάνουμε για τα υπάρχοντα κτίρια και τι εγκαταστάσει. Διότι ε, εάν παραμένουμε στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, απομένουμε στη διάθεση των κρατών μελών για την ανακαίνιση των κτηρίων. Όμω, πρέπει να δούμε το πρόγραμμα σταδιακής δράσης της Επιτροπής, κατά πόσον θα εφαρμοστεί αυστηρά, γιατί δεν είναι βέβαιο κάτι τέτοιο. Και ένα-δυο στοιχεία που μπορεί να μην έχουμε συμπεριλάβει στην έκθεση και πρέπει να τα θυμηθούμε. Λέγαμε παλιότερα ότι όλοι οι τομεί των μεταφορών πρέπει να καλύπτονται από το πρόγραμμα ενεργειακή απόδοση. Να θυμηθούμε εδώ και το θέμα τη χρηματοδότηση που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Διότι Πρέπει να δοθούν περισσότερες δυνατότητες στα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και περισσότερες απαιτήσει για το φάσμα χρηματοδοτικών μέσων που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν. Θέλουμε λοιπόν η έκθεση αυτή πραγματικά να είναι ισχυρή και να επηρεάσει, διότι δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Ε, είμαστε βέβαιοι από τα αποτελέσματα ότι ήδη κάνουμε το μισό των προσπαθειών που απαιτούνται για να πετύχουμε το 20% εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι το 2020. Σε κάθε περίπτωση όμω αυτό που σίγουρα χρειαζόμαστε είναι ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει δράσει. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε η έκθεσή μα να το πετύχει αυτό. Να καταφέρουμε να έχουμε εξοικονόμηση από την πλευρά τη ενεργειακή απόδοση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο Σιμάνσκι. Ε, ευχαριστώ. Όντω. οι εργασίες αυτές ε, και το περιεχόμενο της έκθεσης είναι πολύ σωστές και νομίζω ότι θα υποστηριχθεί από πολλούς βουλευτές. Εμείς ε, έχουμε και νομοθετική και οικονομική υποστήριξη για την ε, συμπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε πολλά σημεία της έκθεσης αναφέρεται αυτό και είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και την ε, βράχη πρόθεσμη δράση γιατί είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε τις καθυστερήσεις. Επίσης, θα πρέπει να προσθέσουμε ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, να γενικεύσουμε το σύστημα των λευκών πιστοποιητικών. Έχω την αίσθηση ότι η μέχρι στιγμής πείρα μας έχει δείξει ότι τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση. Μπορεί μερικές φορές και να διπλασιάσουν τις οικονομίες που γίνονται σε πολλά κράτη-μέλη. Γι' αυτό σε διάφορες νομοθετικές πράξεις καλό θα ήταν να γενικεύσουμε το σύστημα των λευκών πιστοποιητικών. Διαφωνώ όμως με ένα θεμελιώδες θέμα, γιατί ο στόχος αυτής της ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. Διαφωνώ με το δεσμευτικό χαρακτήρα. Ο ενδεικτικός χαρακτήρας είναι καλύτερος, είναι πιο ελαστικός, δίνει περισσότερες δυνατότητες στα κρατημέλη, μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών και δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο που θα εξοικονομήσουν την ενέργειά τους. Ενώ αν έχουμε δεσμευτικούς στόχους, όπως σε άλλες νομοθετικές πράξεις, ούτως ή άλλως δεν έχουμε εγγυήσεις για την υλοποίηση αυτών των δεσμευτικών στόχων. Γιατί μερικές φορές ε, παρόλα αυτά αποτελέσματα δεν λαμβάνουμε ακόμη και με υποχρεωτικούς στόχους. Θα πρέπει να έχουμε ισχυρούς μηχανισμούς ε, παρακολούθησης και ελέγχου. Προτιμώ αυτό το σύστημα ενίσχυσης του ελέγχου γιατί νομίζω ότι έτσι θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα το, στόχο, το βασικό στόχο της έκθεσης. Έχουμε καταθέσει και σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή, ο κύριο Βιντάλ Κουάδρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μπέντσεν για το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμή, αλλά και για αυτό που του έχει απομείνει από εδώ και πέρα. Μαζί με την κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα, ο κύριος Μπέντσεν αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο της αξιολόγησης ε, εδραίωσης αλλά και της χάραξης της μελλοντική μας ενεργειακής πολιτικής σε πολύ χαλεπούς καιρούς γιατί διανύουμε μια πολύ σοβαρή κατάσταση σοβαρο... Ε, δεινής κρίσης. Οι δύο αυτές ε, εκθέσεις είναι αλληλένδετες. Οπότε καλό θα είναι και η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε να είναι συνεπής. Δεν μπορούμε να έχουμε αντιφάσεις στην ε, προσέγγισή μας στις δύο εκθέσεις. Συμφωνώ και με τους δύο εισηγητές ότι είναι κεφαλαιόδου σημασία η σωστή και άμεση εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, της ισχύουσης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και επικροτώ την παράγραφο 5 της έκθεσης Μπένσεν, στην οποία επιμένει στο σημαντικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη στιγμή έναρξης ε, διαδικασιών επί παραβάση κατά των κρατών μελών είναι αναφυσβήτητο ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε σωστά την ισχύουσα νομοθεσία πριν να ε, εμπλακούμε σε νέες περιπέτειες. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας δίνει αυτή η έκθεση και να αξιολογήσουμε εις βάθος και να εδραιώσουμε το ενεργειακό μας κεκτημένο. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν υποβάλουμε νέες πρωτοβουλίες. Επίσης, ε, Συμφωνώ και με την παράγραφο 4 της έκθεσης Μπένσον. Εκεί ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει με κριτικό τρόπο τα εθνικά σχέδια απόδοση και το βαθμό εφαρμογής τους. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να εκτιμήσει την πρόοδο που έχει γίνει με βάση τα μέχρι τώρα μέτρα και να προσδιορίσει καλύτερα τους στόχους της εν της στρατηγικής του 2020. Όλοι έχουμε επίγνωση ότι ακριβώς επειδή δεν υλοποιήσαμε τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, πλήξαμε σοβαρά το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αξιοπιστία της και την δυνατότητά της να προσδιορίσει και να υλοποιήσει διάφορους στόχους. Η θέσπιση δεσμευτικών στόχων δεν θα πρέπει να είναι ε, αιώνια πηγή ματέωσης και απογοήτευσης. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε τους στόχους μας με αποφασιστικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακας της ε, Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και θα πρέπει επιτέλους να ανακτήσουμε τη χαμένη εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου πολίτη και θα πρέπει αυτό να το καταφέρουμε με συγκεκριμένες δράσεις ε, συνεπείς, αποτελεσματικές και απτές και να αποφύγουμε ε, ουτοπικές πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να καταθέσω και ορισμένε τροπολογίε και να σα και το περιεχόμενό τους. Είναι σαφές από αυτά που είπα ότι κατά τη γνώμη μου δεν είναι σήμερα συνετό να προσθέσουμε νέους δεσμευτικούς στόχους στη στρατηγική μας για την ενεργειακή απόδοση. Όταν κάνουμε βεβαιασμένες ενέργειες δεν θα έχουμε αποτελέσματα θετικά. Κάθε κράτος μέλος θα μπορεί αυτόνομα να επιλέξει το τύπο ενέργειας, ενεργειακού μείγματος που θα οδηγήσει σε αξικονόμηση ενέργειας. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την παράγραφο 9, όπου ζητείται προ, προαγωγή της ε, συνδυασμένης παραγωγής για το district heating. έχουμε διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες στο βορρά και στο νότο. Άλλο ε, συμπαραγωγή στο βορρά και άλλο στο νότο. Δεν μπορούμε λοιπόν να προβαίνουμε σε διακριτική μεταχείριση των διαφορετικών τρόπων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι πριν από λίγα χρόνια, το 2006, είχα συντάξει μια έκθεση πρωτοβουλίας για την ενεργειακή απόδοση και για τα περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα. Εκεί είχα επιμείνει στο άλλο πράγμα είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης που είναι πολύ καλό και άλλο μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό είναι επικίνδυνο γιατί ιδιαίτερα σε εποχές ύφεσης δεν μπορούμε να θέτουμε σε κίνδυνο την οικονομική μας ανάπτυξη. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτές τις έννοιες. Γι' αυτό και θα καταθέσω σχετική τροπολογία. Αυτά κύριε Πρόεδρε και ευελπιστώ ότι αύριο, μετά από αυτή την καρποφόρα συζήτηση που είχαμε, θα συνεχίσουμε το δρόμο προς τη διαμόρφωση ενός ισορροπημένου κειμένου που θα τύχει της ευρύτερης δυνατής υποστήριξης. Ο κύριος Τσουκαλάς. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Μπέντσεν για την πολύ καλή δουλειά του και να επισημάνω ορισμένα πράγματα. Η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που μπορεί να οδηγήσει σε ένα εντελώς καινούριο οικονομικό και ενεργειακό μοντέλο. Και σε αυτή τη μετάβαση οι τεχνολογίες που αναπτύσσονται σήμερα και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως οι νανοτεχνολογίες ή η φωτονική, μπορούν να παίξουν μείζωνα ρόλο. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών οφείλουν να χρησιμοποιηθούν έξυπνα για την προώθηση μιας πιο συνειδητής ενεργειακής κατανάλωσης τόσο στα νοικοκυριά και στις μεταφορές, όσο και στην παραγωγή ενέργειας και στη βιομηχανία. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας του ίδιου του τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως σε εκθέσεις μας εδώ έχουμε ζητήσει. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας στους λεγόμενους έξυπνους μετρητές. Οι έξυπνοι μετρητές διαθέτουν ένα τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Μόνο όμως η Ιταλία, Σουηδία και Φιλανδία αγγίζουν το 100% της διείδησης των έξυπνων μετρητών. Άλλα κράτη-μέλη όμως βρίσκονται αρκετά πίσω μόλις στην φάση εκπόνησης μελετών για τη δυνατότητα εφαρμογής των έξυπνων μετρητών. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε εγκαίρως είναι ένα σαφή πανευρωπαϊκό ορισμό του τι ακριβώς είναι ένα smart meter και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξή τους. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι έξυπνοι μετρητές επιφέρουν αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών ενέργειας μόνο όταν τους ενημερώνουν για την κατανάλωσή τους, δηλαδή διαθέτουν οθόνες ή ο χρήστης μπορεί μέσω του διαδικτύου να συνδεθεί και να δει λεπτομέρειες για την κατανάλωσή του. Στόχος μας πρέπει να είναι και η ενημέρωση των καταναλωτών και όχι μόνο η εξυπηρέτηση των παρόχων για αυτοματοποιημένες και φθηνές τηλεμετρήσεις της κατανάλωσης. Όσο για το χρονοδιάγραμμα, ας μην ξεχνάμε ότι στην έκθεση της κυρίας Δεκαστήγιο για την ψηφιακή ατζέντα ταχθήκαμε υπέρ του στόχου 50% των οικοκυριών να είναι εξοπλισμένα με έξυπνους μετρητές ως το 2015. Βέβαια, δεν αρκούν οι έξυπνοι μετρητές αναγκαία είναι και η ανάπτυξη έξυπνων συσκευών συμβατών με τους έξυπνους μετρητές που θα προσαρμόζονται αυτόματα στα επίπεδα κατανάλωσης και τις ανάγκες των ενεργειακών δικτύων. Τέλος, με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην έκθεση γίνεται αναφορά και στον ηγετικό ρόλο που οφείλουν να διαδραματίσουν τα κτίρια των ευρωπαϊκών οργανισμών στη μετάβαση σε κτίρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2020. Και πάλι με τα συγχαρητήρια σας ευχαριστώ. Next, next Wortmeldung ist Kollegin Hübner. Thank you very much, Mr. Chairman. Hey, ναι, um, excuse me. Συγγνώμη, η συνάδελφος Χίπνερ, λέει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Ε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και ευχαριστώ θερμά για όλες τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν για το θέμα αυτό. Σήμερα, συνάδελφοι, μιλούμε για ένα εξαιρετική σημασία ζήτημα για ένα σπουδαίο θέμα, όχι μόνο για την πολιτική μας ως προς το κλίμα και την περιβαλλοντική μας πολιτική, αλλά και για τα οικονομικά προβλήματα που έχουμε σε πολλές χώρες. Η εξορθολόγηση της χρήσης, ο εξορθολογισμός της χρήσης ενέργειας θα πρέπει να είναι εξίσου σημαντική προτεραιότητα, όπως και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, και οι επενδύσει σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ε, είναι σημαντική, όπω και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και η εξοικονόμηση τη ενέργεια, η ενίσχυση τη ενεργειακή απόδοση, που δυστυχώ δεν είναι ακόμη καλά προσδιορισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική η συγκεκριμένη έκθεση. Γι' αυτό είναι σημαντική η απόδοση τη ε, δέουσα προσοχή στο θέμα τη ε, ενεργειακή απόδοση. Όταν μιλούμε για εξοικονόμηση ενέργεια, ε, ας μην ξεχνούμε ότι είναι απαραίτητο αυτό για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών μας στόχων. Γιατί η αγορά από μόνη της δεν καταφέρνει να ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιες ε, ενέργειες από πλευράς χωρών. Χρειάζεται ρύθμιση και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η εξοικονόμηση της ενέργειας μας χρειάζεται, μας είναι απαραίτητη για να ε, αναγκάσουμε τον καταναλωτή να κάνει μια πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας, αλλά το ίδιο και τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει και οι επιχειρήσεις να κάνουν εξοικονομήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς πόρο απέχει από τις Ηνωμένε Πολιτείε ή από την Ιαπωνία σε τα θέματα αυτά της απόδοσης. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία για μας αυτό το θέμα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξοικονόμησης της ενέργειας. Όπως ανέφερα και συνάδελφοι, έξυπνοι μετρητές, αλλά και το θέμα της, του φωτισμού των δρόμων, για παράδειγμα. Γιατί εκεί χάνουμε πολύ ενέργεια με το φωτισμό θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το θέμα με μεθόδους ε, μεγαλύτερης εξοικονόμησης ενέργειας. Θα πρέπει να δούμε και τι ενεργειακή κατανάλωση έχουν συγκεκριμένα προϊόντα. Γι' αυτό και χρειάζονται εκστρατείες ε, για καλύτερη ενημέρωση. Χρειάζεται επιμόρφωση και των εργαζομένων στον ενεργειακό κλάδο έχουμε ισχύουσες διατάξεις για την ανακαίνιση των κτηρίων υπό το πρίσμα της ενεργειακής τους απόδοσης. Αυτό το θέμα είναι σημαντικό και υπάρχουν όπω είπα σχετικέ διατάξει, αλλά δυστυχώ στην πράξη δεν έχουμε τους σωστή εφαρμογή. Για παράδειγμα, πολλά κτίρια δεν α, τηρούν αυτές τις προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης. Βέβαια, θα πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων, όχι να τιμωρήσουμε τους μεν ή τους δε. Για παράδειγμα, θα πρέπει να προωθήσουμε ε, προϊόντα που δεν είναι ενεργειοβόρα. Θα πρέπει να δώσουμε ενάψματα και να ενθαρρύνουμε αυτούς ε, που επενδύουν, επενδύουν στις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη διαφοροποίηση των διαφόρων πηγών ενέργειας. Τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης θα είναι σημαντικά όχι μόνο για την περιβαλλοντική προστασία, αλλά θα συμβάλλουν και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, γιατί ε, αυτό το θέμα είναι επίσης σημαντικό. Επίσης, ε, η βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εξίσου είναι σημαντικό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται ως πρωταγωνιστής, ε, διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο θέμα της χρήσης φιλοπεριβαλλοντικής ενέργειας. Επίσης, δίνουμε ε, μάχη για να μειώσουμε σε σχετικά μικρό ορίζοντα μέχρι και 80 με 95% τις εκπομπές του άνθρακα και θα πρέπει να γενικεύσουμε τις προσπάθειες για την εξορθολόγηση της ε, ε, ενεργειακής κατανάλωσης. Βέβαια, η πολιτική αυτή δεν θα πρέπει να έχει βραχυπρόθεσμο ή κοντόφθαλμο στόχο. Θα πρέπει να έχουμε και μία πιο μακροπρόθεσμη προοπτική αν ε, αυξήσουμε τις δαπάνες μας στα θέματα εξορθολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης, τα αποτελέσματα θα είναι θετικά όχι μόνο για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε στόχους και στην παγκόσμια κοινότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γκέρεκ. Ε, Ευχαριστώ. Η ενέργεια δεν καταναλώνεται μόνο, γιατί φαίνεται να μιλούμε μόνο για την κατανάλωση, μιλούμε ω καταναλωτέ. Δυστυχώ πολλά στοιχεία λείπουν από την έκθεση. Η ενέργεια δεν είναι ε, προϊόν της αγοράς, δεν υπόκειται σε καταστροφή. Καλύτερα να μιλούμε για χρήση της ενέργειας, όχι κατανάλωση ενέργειας, γιατί η ενέργεια δεν αναλώνεται. Επίσης ε, θέλουμε όλος, όσο δυνατόν περισσότερη αποτελεσματικότητα όταν μιλούμε για αποτελεσματικότητα, είναι σαν να μιλούμε για φυσικοχημικές πτυχές. Ε, πριν όμως την, ε, ε, τη φάση της αγοράς. Μιλούμε επίσης για οικονομικές πτυχές, όπως είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης, γιατί αυτό φαίνεται ότι τονίσαμε περισσότερο στη συζήτηση. Σίγουρα θα πρέπει να επιβάλλουν ένα εξορθολογισμό της κατανάλωσης, αλλά αυτό δεν γίνεται ξεχωριστά από μια ανεξάρτητη οργάνωση. Νομίζω ότι οι βασικές δυνατότητες για την ε, εξοικονόμηση βρίσκονται στο στη φάση της ε, την φυσικοχημική, της αλλαγής, ε, της μετάβασης από ένα τρόπο ενέργειας στο, σε άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, έχουμε διάφορες μορφές ενέργειας, ατομική, άνθρακα, αυτό είναι όμως ε, περισσότερο ε, εξοικονόμηση της ενέργειας και σχεδιασμός της ενέργειας σε φάση πριν ε, την αγορά. Και οι περισσότερες εξοικονομήσεις μπορούν να γίνουν σε αυτή τη φάση. Έχουμε πολλές φορές απώλειες στα δίκτυα της ενέργειας. Γιατί δεν αναφέρεται τίποτα τέτοιο στην έκθεση στη χημεία στις, ε, ή στις, ε, στους πυρηνικούς σταθμούς έχουμε τεράστιες απώλειες πηγές ενέργειας. Γιατί δεν ναι. μιλούμε για την ενεργειακή απόδοση και εκεί. Η ενεργειακή απόδοση στους πυρηνικούς σταθμούς είναι πολύ λιγότερη από την ενεργειακή απόδοση των ε, ε ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών με άνθρακα. η θερμοαπομόνωση, πολύ σωστά πρέπει να αναφέρεται. Επίσης ε, υπάρχουν πολλοί, μηχανικοί τρόποι και τεχνικοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας που δεν αναφέρονται στην έκθεση. Για, τις, ε, για τα μαγνητικά πεδία υπάρχουν ε, μερικοί μερικά εργοστάσια που μέχρι και 2% χάνουν την αποτελεσματικότητά τους εξαιτίας κακής χρήσης των μαγνητικών πεδίων. Έχουμε φυσικό αέριο. Από το φυσικό αέριο παράγουμε θερμότητα. Από τη θερμότητα παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Στέλνουμε το ηλεκτρικό ρεύμα στον ε, καταναλωτή και το χρησιμοποιεί για θέρμανση. Έχουμε ελάχιστη αποτελεσματικότητα. Στην αλυσίδα αυτή ξεχνούμε τελείως το κλάδο της μετατροπής. Και δυστυχώς από τη μετατροπή, από τη μία πηγή ενέργεια στην άλλη είναι που έχουμε τεράστιες απώλειες στην ενέργεια. Θα πρέπει την ενεργειακή απόδοση να την ε, εντοπίσουμε στη χρήση και όχι στην κατανάλωση. Γιατί και το θέμα της ε, εντροπίας στο περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό, αλλά αυτό είναι θέμα που απασχολεί περισσότερο τους περιβαλλοντολόγους. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά του, τον συνάδελφο Μπέντσεν, και κυρίω για τη μέθοδο που ακολούθησε για την σύνταξη αυτή τη έκθεση. Πραγματικά προσυπογράφουμε στα περισσότερα σημεία. Κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι έχουμε πολλέ ε, πιθανότητες και λόγω της κοινωνική κρίσης και λόγω της οικονομική κρίση που διανύουμε το δυναμικό μας της δημιουργίας απασχόλησης, το δυναμικό του δικτύου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μην γίνεται αρκετά γνωστό προς τους πολίτες μας ώστε να χρησιμοποιείται για σκοπούς ενεργειακής απόδοσης. Αντιθέτως, αυτό που δεν θα μας συγχωρήσουν οι συμπολίτε μας είναι όταν το βαρέλι θα φτάσει, το πετρελαίο θα φτάσει πάλι τα 150 δολάρια, να μην έχουμε εμείς ε, προβλέψει τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό που διαθέτουμε για εξοικονόμηση ενέργεια. Διότι θα είναι εκείνη τα πρωταθήματα τη επόμενη ενεργειακή κρίση. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε στο τέλο του χρόνου και εδώ θα συμφωνήσω με τα σχόλια που έγιναν περί χρονοδιαγράμματο, πρέπει οπωσδήποτε στο τέλο του χρόνου να έχουμε ένα πραγματικό πρόγραμμα δράση για την ενεργειακή απόδοση. Όχι μόνο με λόγια και ωραίε εκφράσει, αλλά με συγκεκριμένε προτάσει, συγκεκριμένα μέτρα ε, αναθεώρηση οδηγιών, στόχους ποσοτικούς και ποιοτικούς που να διευκρινίζονται επακριβώς στο σχέδιο. Βεβαίω θέλουμε να υπάρχουν στόχοι δεσμευτικοί. Χθε μάλιστα συζητήσαμε το θέμα των αγωγών. Των αγωγών φυσικού αερίου, είτε είναι ο Ναμπούκο, το South Stream ή το North Stream. 20% ε, της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη ισοδυναμεί με 15 αγωγούς σαν τον Ναμπούκο. Το 20% λοιπόν, όπως είπα, της ενεργειακής απόδοσης στην Ευρώπη ισοδυναμεί με 15 ναμπούκους, 15 ναφουγοδονόσορες. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό. Και είναι και πολύ πιο φτηνό να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό που είναι μια πραγματική λεωφόρο προ την ε, ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργεια. Ω προ το περιεχόμενο τη έκθεση, συμφωνώ με του περισσότερου στόχου που διατυπώνονται από τον εισηγητή και πιστεύω ότι για την ανακαίνιση των υπαρχόντων κτηρίων θα πρέπει να θέσουμε πραγματικά την προτεραιότητα όπως και ο εισηγητής σε αυτόν τον τομέα. Οι πρωτοβουλίε, οι σχετικέ, ο ρυθμό ανακαίνιση των κτηρίων, η ποιότητα τη ανακαίνιση, νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, να είμαστε πιο φιλόδοξοι, γιατί υπάρχει μεγάλο δυναμικό από την άποψη τη εξοικονόμηση τη ενέργεια ως προς την ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα που σήμερα υποφέρει από οικονομικής άποψης. Και μάλιστα σοβαρά. Για την θεματοδότηση, είναι και αυτό κέρια σημασία ζήτημα, και πάλι ο εισηγητή φαίνεται να του δίνει τη σωστή σημασία. Οδεύει προ τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι με τι τροπολογίε μας για το θέμα αυτό θα μπορούσαμε να ζητήσουμε επιπλέον από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν την υποχρέωση να υλοποιούν σε κάθε χώρα τα σχετικά ένα ταμείο ενεργειακής απόδοσης που θα χρησιμοποιεί κάποια κονδύλια δημόσια και ένα μέρος ιδιωτικών κονδυλίων. Τι ερχόμενε εβδομάδες θα έχουμε συζητήσει για την οδηγία της ενεργειακής φορολογίας, τη φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και βεβαίω θα αρχίσουν να δημοπρατούνται και οι ποσοστώσει ε, διοξιδίου του άνθρακα βάσει τη σχετική οδηγία. Εδώ μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την ενεργειακή απόδοση από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν πολλέ πηγέ. Και υπάρχουν πολλά ορυκτά καύσιμα και κατανάλωση ορυκτών καυσίμων περιττή και πολύ dumping ε, για την κατανάλωση ενέργεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεκάδε δισεκατομμύρια επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα ή για την συμπαραγωγή. Εδώ λοιπόν πρέπει να φανούμε συνεπείς προ τα πολιτικά μας μέτρα και ω προς την ποιότητα της ενεργειακής απόδοσης. Προφανώς, εάν έχουμε στόχους φιλόδοξους και δεσμευτικούς για την εξοικονόμηση ενέργειας, οι πλέον ευάλωτοι πληθυσμοί στην Ευρώπη θα είναι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν. Ω προ την αγοραστική του μάλιστα δύναμη. Όμω χρειαζόμαστε και συγκεκριμένα εργαλεία. Και επειδή δεν γίνονται αρκετά στα κράτη-μέλη, να άλλο ένα τομέα όπου υπάρχει ευρωπαϊκή ευθύνη. Να αναλάβουμε το θέμα αυτό τη ε, επισφαλού ε, ενεργική κατάσταση. Thank you very much, Καρβάλιο. Uh, uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε, να συγχαρώ τον κύριο Μπένσεν για την πολύ καλή του έκθεση και για την ισορροπία που πετυχαίνει μεταξύ των ε, σημερινών οικονομικών περιορισμών και των φιλοδοξιών για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Ε, σε αυτό το σκηνικό θα πρέπει να αναζητήσουμε νέους τρόπους για να δώσουμε κίνητρα προκειμένου να πετύχουμε ενεργειακή απόδοση και μια δυνατότητα που θα ήθελα και εγώ να προτείνω, με τροπολογία που ήδη συζητήσαμε και με τον ίδιο τον εισηγητή, είναι να προβλέψουμε την ιδέα της ε, ε, επιβολής κριτηρίων για την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δηλαδή, τα προγράμματα θα χρηματοδοτούνται, αυτή τη στιγμή πετυχαίνουν κάποιε προδιαγραφέ, κάποια πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση. Δεν θέλουμε πολύ δαπανηρά, πολύ ακριβά προγράμματα για, ανανεργε... για ανανεώσιμε ενέργειε με χρήση λόγω χάρη εάν το κτίριο τελικά δεν είναι ε, από ενεργή άποψη αποδοτικό. Εκεί θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση λοιπόν και προ τα εκεί να προωθήσουμε την ενεργειακή απόδοση στο μέλλον. Έπειτα, είναι πολύ σημαντικό σε επίπεδο δημοτικών αρχών και τοπικών αρχών να αναλυθεί δράση. Η Ευρώπη έχει ένα ολόκληρο δίκτυο φορέων και οργανισμών που έχουν δημιουργηθεί με ευρωπαϊκή στήριξη και ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι δημοτικές και τοπικές αρχές, φορείς υπεύθυνοι για την ενέργεια, μπορούν να αναφέρονται και στην έκθεση, πιστεύω. Και τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε το ρόλο της ε, βιομηχανίας εδώ σε αυτόν τον τομέα, ιδίω από την πλευρά τη έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών. Κατά την έποψη μου, η βιομηχανία που από τεχνολογική άποψη λειτουργεί πολύ εντατικά πρέπει να κάνει περισσότερη έρευνα και να αναζητήσει περισσότερη τεχνολογική ανάπτυξη. Υπάρχει ανάγκη να αναζητηθούν νέε, ανανεωμένε διαδικασίε σε κάποιου τομεί τη βιομηχανία, προκειμένου να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί και στο μέλλον. Εξασφαλίζοντα ενεργειακή Επιτρέποντα μάλλον να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια και να αντιμετωπίζουμε του περιβαλλοντικού μα περιορισμού. Να λοιπόν ποια είναι η σημασία τη έρευνα για την εξοικονόμηση ενέργεια στη βιομηχανία με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή, ενεργειακά εντατική βιομηχανία. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ από πλευρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή και να τον συγχαρώ. Θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες κι εμείς. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω ότι θεωρώ ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί, θα πρέπει να αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον. Πιστεύω και ελπίζω η ενεργειακή αποδοτικότητα να μπει τόσο στην ατζέντα του Συμβουλίου όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την ενεργειακή ένδυα τώρα, όπως ε, ανέφεραν και οι συνάδελφοι, ο αριθμός των όσων πλήττονται από την οικονομική αυξήθηκε λόγω κρίσης κάτι την οικονομική ύφεση. Γι' αυτό όλο και πιο πολλές οικογένειες στην Ευρώπη πλήττονται από την ενεργειακή ένδια. Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος αυτού, όπως ε, Ζήτησα και στην έκθεση για την αποδοτικότητα των κτηρίων, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων, θεωρώ. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα περιφερειακά ταμεία, προκειμένου τα σχέδια που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων να έχουν πιο υψηλή προτεραιότητα. Προτείναμε το 4%. Ελπίζουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά και τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές προκειμένου να τονίσουμε ιδιαίτερα τη σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων. Επίσης, τέθηκε το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας της μεταφοράς. Ναι. Είναι σωστό και η σχετική σύσταση προς την κατεύθυνση αυτή για τη βελτίωση τη ενεργειακή αποδοτικότητα και στον τομέα των μεταφορών. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα. που απευθύνονται στην εντατικοποίηση των τομέα των μεταφορών. Και εδώ παρουσιάζονται η ανάγκη να κοιτάξουμε και τα ηλεκτρικά μηχανήματα. Μπορούμε να μιλήσουμε και για ποδήλατα. Οι συσκευές αυτές λοιπόν θα πρέπει να συνδέονται ίσως με ευφυή e συστήματα, δίκτυα. Ελπίζω να με ακούει και ο εισηγητής. Η χρήση των ανεώσιμων έχει μεγάλο δυναμικό και το πρόβλημα που παρουσιάζεται σήμερα είναι για παράδειγμα ότι στην, Γερμανία, στην Ισπανία δαπανώνται 5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τι ανανεώσιμε ε, πηγές και ουσιαστικά αυτές οι επενδύσεις πήγαν χαμένες γιατί δεν υπάρχει το δίκτυο για την αξιοποίηση της ενέργειας αυτής. Όταν αναπτύσσεται λοιπόν η υποδομή θα πρέπει να, γίνει αυτό, να γίνεται αυτό σε τοπικό επίπεδο προκειμένου αυτές οι ηλεκτρικές συσκευές να είναι δυνατόν να ενσωματωθούν σε ένα ευφυές δίκτυο. Κλείνοντας, να αναφέρω το εξή. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων, δεν έχουμε καταφέρει όλα όσα θέλαμε και περιμένουμε περαιτέρω έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και η παρέτητη χρηματοδότηση προ την κατεύθυνση αυτή. Ο συνάδελφο Ευχαριστώ, Νομίζω ότι αναφυσβήτητο ότι η ενεργειακή απόδοση είναι σημαντική για την ανταγωνιστικότητα, για την ασφάλεια, αλλά και για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών πηγών. Γιατί εξορθολογίζοντας ε, και κάνοντας πιο αποτελεσματική τη χρήση της ενέργειας, είναι πιο εύκολο να περάσουμε και σε νέες πηγές ενέργειας. Νομίζω ότι ένα σημείο θα πρέπει να το τονίσουμε στην έκθεση, και ευχαριστώ τον ε, εισηγητή που το κάνει ήδη. Το θέμα είναι ότι όταν αναλαμβάνουμε κάποιες δράσεις θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι για τα νοικοκυριά, για τους ιδιώτες, για τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε συμφέρον ε, να εξορθολογήσουμε τη χρήση ενέργειας εξαιτία των υψηλών τιμών της ενέργειας. Θα πρέπει όμως να δώσουμε έμφαση στους τομείς όπου εμείς ή είτε ως επιχειρήσει είτε ως πολίτες δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η ενέργεια. Εμείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις διάφορες δημόσιες δομές. Για παράδειγμα, αναφέρεται η στέγαση, η, συγγνώμη, η θέρμανση στις πόλεις, η, το θέμα της ενέργειας στις μεταφορές. Γιατί όταν μιλούμε για δεσμευτικούς υποχρεωτικούς στόχους, νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιούμε δεσμευτικές δράσεις όταν υιοθετούμε μια μεγαλύτερη προοπτική και πιο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το θέμα της στέγασης των σπιτιών ή το θέμα της ενέργειας της μεταφορές. Αυτή την προσέγγιση θα τονίσω με τις τροπολογίες μου. Και όσο πιο ανήμποροι είναι οι ιδιώτες να επηρεάσουν τα πράγματα, τόσο πιο επιτακτική θα είναι ανάγκη να υποβάλουμε κάποια μέτρα σε επίπεδα ένωσης. Ο κύριος Μπρεζίνα. Ευχαριστήσουμε τον εισηγητή. Γιατί όλε οι προτάσει είναι ιδιαίτερα θετικέ. Οι δεσμευτικοί στόχοι θεωρώ ότι είναι σημαντική αν και είναι λίγο νωρί για να είναι δεσμευτική. Όμω, όσο καλύτερα χρησιμοποιούμε την ενέργεια, τόσο καλύτερα θα λειτουργούν και τα συστήματα διανομή μα και όλα θα είναι καλύτερα έτσι. Εάν διασφαλίσουμε την ενεργειακή βεβαιότητα, ασφάλεια, καλύτερη, θα, η Ευρώπη θα δίνει καλύτερη εικόνα. Θα είναι θετικέ οι συνέπειε για ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Ωστόσο, Εδώ ίσως φάλουμε. Μπορεί να κάνουμε ένα τεράστιο σφάλμα. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας, να μην χρησιμοποιούμε τόση ενέργεια σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Όμως το να κινητοποιήσουμε ολόκληρη την κοινωνία, αλλάζοντας επιμέρους ε, νόμους και κανόνες, δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε αν δεν είμαστε εμπειρογνώμονες. Υπάρχουν και οικονομικές ανάγκες και προτεραιότητες. Και αυτό δεν μπορούμε να το παραμελούμε. Με την γενική μείωση της κατανάλωσης δεν σημαίνει ότι θα άμεσα θα πετύχουμε και ενεργειακή απόδοση. Δηλαδή, τα, οι λάμπες που χρησιμοποιούνται και είναι, ε, είναι, πιο, είναι ενεργειακά αποδοτικότερες, αν αυτές αντικατασταθούν και αντικαταστήσουν τις παλιές, δεν σημαίνει ότι θα πετύχουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, διότι μπορεί να χρησιμοποιούνται περισσότερες λάμπες τελικά. Άρα να υπάρξει επίπτωση και σε οικονομικό επίπεδο. Για όλες λοιπόν τις προτάσεις συμφωνώ πέραν των δεσμευτικών στόχων. Αυτή είναι η μόνη εξαίρεση. Συμφωνώ με την ε, φιλοδοξία της ενεργειακής απόδοσης, αλλά μην πιστεύουμε ότι με την ενεργειακή απόδοση μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες εξοικονομήσεις ενέργειας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Δύο θέματα είναι που με προβληματίζουν. Καταρχήν θα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Έκανε τεράστια προσπάθεια για να παραμείνει ρεαλιστής. Γιατί υπάρχουν πολλά θέματα στο ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης. Πολλές φορές ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιφατική. Δεν μπορούμε να μιλούμε κάθε μέρα για την οικονομική κρίση και να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα για τα θέματα ενεργειακής απόδοσης. Στην Ισπανία έχουμε περίπου 5 εκατομμύρια ανέργους. Μόνο το 1% από αυτούς μπορούν να αλλάξουν αυτοκίνητο. Και ποιος μπορεί να ανακαινήσει το σπίτι του. Μπορεί και κανένας. Το κόστος του ηλεκτρισμού στην Ισπανία, του ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήθηκε κατά 60%. Φανταστείτε λοιπόν, τι κόστος έχουν οι επιχειρήσεις. Και όλα αυτά επειδή δεν έχουμε πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ πιο δαπανηρές. Είναι αντιφάση, υποπίπτουμε συνεχώς σε αντιφάσεις. Γιατί μιλούμε για τη φτώχεια, μιλούμε για την ισότητα, αλλά ταυτόχρονα επιβαρύνουμε τους φτωχούς με όλο και μεγαλύτερο άχθος και με όλο και μεγαλύτερα έξοδα. Επίσης, μιλούμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα επιτρέψουν ε, στους Δήμους ένα είδος αυτονομίας. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, μας υποχρεώνουν να μιλούμε για τα μεγάλα ηλεκτρικά δίκτυα που μεταφέρουν ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε εμείς ε, στην Καρταχένα από την Νότια Ισπανία να εφοδιάζουμε την Καταλωνία με ρεύμα. Μια λέμε μαύρο, μια λέμε άσπρο. Συνέχεια φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Και αυτή η τακτική με προβληματίζει ιδιαίτερα. Γιατί σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την εκτίμηση των επιπτώσεων και για τον οικονομικό αντίκτυπο. Αν όμως θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι, θα πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση, μια αξιολόγηση των επιπτώσεων των αποφάσεών μας γιατί φαίνεται ότι εμείς είμαστε αριστοκράτες και περιφρονούμε πλήρως την Επιτροπή των Περιφερειών και τους Δήμους, γιατί εμείς μπορεί να χαράζουμε τους νόμους, αλλά αυτοί που τους εφαρμόζουν είναι οι Δήμοι και οι κοινότητες και δεν τους διευκολύνουμε καθόλου. Όλο αντιφάσεις είμαστε. Συμφωνώ με τον εισηγητή, γιατί με αυτό το binding, αυτούς τους δεσμευτικούς στόχους, ε, θέλουμε στόχους ώστε να μπορούν και οι 5 εκατομμύρια άνεργοι να ανακαινήσουν το σπίτι τους και να μην πρέπει να ε, πληρώνουν και πρόστιμο αν δεν μπορούν να το κάνουν. Σε ό,τι αφορά την ε, οικολογική ετικέτα, η ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία είναι τόσο καινοτόμα που αν ε, επιβάλα, αν έπρεπε να επιβάλλουμε οικολογική ετικέτα σε όλα τα προϊόντα, θα σταματούσαμε την καινοτομία. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάζουμε. Η διοίκηση δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάζει ετικέτες κάθε, κάθε δύο χρόνια. Η καινοτομία όμως και η τεχνολογία προχωρούν με ραγδαίους ρυθμούς, πολύ πιο ραγδαίους από τους ε, ρυθμούς της διοίκηση. Δεν μπορούμε να υποτάξουμε την καινοτομία στον βραδύ ρυθμό της διοίκηση. και αυτό θα κάνουμε με τέτοιες ε, προδιαγραφές. Επίσης, ε, τα, τα μνημεία, τα διατηρητέα. Είναι τα πιο και τα διατηρητέα σπίτια. Είναι τα πιο όμορφα και όμως είναι τα πιο δύσκολα στην αναπαλαίωσή τους και στη συντήρησή τους. Εγώ πρότεινα στην Επιτροπή ένα πειραματικό πρόγραμμα για να δούμε τι κάνουμε για τα ιστορικά κέντρα των πόλεων σε ορισμένε πόλει, όπω ε, σε πόλεις τη Αυστρία. Παρ' όλα αυτά, απορρίφθηκε το, το, η πρότασή μου για το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Όλο αντιφάσει, λοιπόν είμαστε. Από τη μια θέλουμε να υποστηρίξουμε ορισμένα πράγματα και από την άλλη με τις δράσεις μας ουσιαστικά τα υπονομεύουμε. Λυπάμαι που ήμουν τόσο αρνητική, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Να, να προσπαθήσουμε να σας καθησυχάσουμε. Η κυρία Χέτσοκ, η επόμενη μιλητρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας ε, να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή και να πω ότι δεν θα έπαιρνα το λόγο αν είχε υποθεί το πιο σημαντικό το οποίο λείπει, θεωρώ. Η ενεργή αποδοτικότητα είναι ένα ανθρώπινο θέμα. Μιλάμε για ανθρώπους. ο κόσμος μπορεί να την εφαρμόσει όταν ξέρει πώς να την εφαρμόζει. Άρα είναι ένας ε, ορισμένος αναλφαβητισμός, αν θέλετε, ως προς την ενέργεια, ο οποίος επικρατεί. Όταν μιλάμε για την Ήπεθρο, αναρωτιέμαι πόσοι γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει και θα πρέπει λοιπόν αυτό να αποτελέσει πρώτη στην προτεραιότητα από πλευρά παραγωγή να δούμε τι γίνεται, αλλά και από πλευρά καταναλωτή. Θα υποβάλω λοιπόν σχετικές τροπολογίες, μια-δυο, να δούμε και να έχουμε επαφή με τον ηλεκτρολόγο, με αυτούς που χτίζουν τα σπίτια Με αυτόν τον κόσμο θέλουμε επαφή. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε και να περιγράψουμε καλύτερα αυτή την προσέγγιση. Από πάνω προς τα κάτω. Ιδάλλως δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτά ήθελα λοιπόν να αναφέρω εν συντομία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. Θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Η αρμόδια κυρία. Έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, uh, thank you. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπένσεν και όλα τα μέλη που παρενέβησαν από τη δική μας την οπτική ε, γωνία. Η συζήτηση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Είχαμε μεγάλη ανάγκη να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις και μάλιστα πολλές και διαφορετικές απόψεις. Αυτό που πραγματικά είναι ενθαρρυντικό είναι ότι όλοι τόνισαν τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και την ε, σημασία του νέου προγράμματος δράσης της Επιτροπής θα υποβληθεί σύντομα. Είναι ένα καλό σημείο αφετηρία αυτό. Και εδώ αναφέρθηκαν διαφορετικά στοιχεία. Πολλά από αυτά έχουν ήδη συμπεριληφθεί από τον κύριο Μπένσον στην εκθεσή του. Αξιόλογα τα περισσότερα και η Επιτροπή σας διαβεβαιώ ότι θα μελετήσει διεξοδικά όλες τις πρωτοβουλίες και τις ενδείξεις που αναφέρατε θα ξέρετε ότι ένα πρώτο βήμα για να ορίσουμε μια κατεύθυνση πολιτική για το μέλλον της ενεργειακής απόδοσης και το πλαίσιο της είναι η ενεργειακή στρατηγική του 2020. Για το 2020 μάλλον. Οι ευρωπαϊκές ενεργειακές πολιτικές πρέπει να ξεκινήσουν λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της προσφοράς και κατανάλωσης της ενέργειας σε μια πρώτη φάση. Αυτό θα καθορίσει λοιπόν και το πώς θα διαμορφωθούν τα πολιτικού περιεχομένου έγγραφα που θα ακολουθήσουν. Δεν θέλω να, να σταθώ στα λεπτομέρειες που αναφέρθηκαν εδώ. Διότι ούτω ή άλλω θα δούμε το τι συζητήθηκε στην Επιτροπή σα στην τελική μορφή τη έκθεση, όπου θα αντικατοπτρίζονται οι απόψει. Ένα στοιχείο όμω είναι πολύ σημαντικό και αυτό θέλω να το σχολιάσω. Η Επιτροπή καταβάλει σοβαρές προσπάθειες γι' αυτό και άκουσα και κάποιους να το αναφέρουν, να ζητούν αποτίμηση του ισχύοντος πολιτικού πλαισίου. Ξέρετε ότι υπάρχει από το 2006 ένα διεξοδικό σύστημα υποβολής εκθέσεων βάσει του υπάρχοντος πολιτικού μας χαρτοφυλακίου. Αυτό το έργο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, θα εξακολουθήσει και σκοπεύουμε μάλιστα να περατώσουμε και μία ε, συνολική αποτίμηση του πλαισίου αυτού του 2006. Να ένα πρώτο βήμα για να ακολουθήσουν και περαιτέρω πρωτοβουλίες. Εδώ εννοείται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπωσδήποτε θέλει να βεβαιωθεί ότι οι υπάρχουσες πολιτικές πρωτοβουλίες, η υφιστάμενη νομοθεσία και θα προωθηθούν και θα υλοποιηθούν ακόμη πιο εντατικά από τα κράτη-μέλη. Βεβαίως, υπάρχουν σχόλια για τις νομικές διαδικασίες, όμως σημασία έχουν και τα εθνικά προγράμματα για την ενεργειακή απόδοση. Και σε αυτά πρέπει να δοθεί έμφαση. Πρόεδρε, εάν μου επιτρέπετε, εδώ θα ολοκληρώσω η Επιτροπή με τα χαράς να συνεισφέρει και άλλο σε αυτήν την ε, συζήτηση. Και πραγματικά ανυπομονούμε να δούμε το τελικό σχέδιο της έκθεσής σας. Ευχαριστώ. Μία μικρή υπόδειξη για την υπόλοιπη συζήτηση. Ελπίζω να μην κατάλαβα σωστά. Είπατε η βάση για τις περαιτέρω διαβουλεύσεις ποια θα είναι. Δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε τώρα, αλλά φαντάζομαι ότι θα ενημερωθούν τα έγγραφα αυτά. Το 2006 δεν μπορεί να είναι πραγματικά το έτος αξιολόγησης των όσων ε, έγιναν, αλλά να δώσω το λόγο στον κύριο Μπέντσεν για να μας απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Όχι, δεν είναι δίκαιο αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχήν όλους και οδησηγητές αλλά και τους υπόλοιπους συναδέρφους για τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους. Είχαμε συζήτηση για την ενεργειακή ένδυα, την παιδεία, τις μεταφορές αλλά και το στόχο της ανακαίνησης των κτηρίων. Όλα τα σχόλια ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Και όπως είπα, χρησιμοποιούμε πολύ από την ενέργειά μας στα παλιά κτίρια. Και η οδηγία για την ανακαίνιση, ή η οδηγία μάλλον για την ενεργειακή απόδοση αφορά τα νέα κτίρια. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να καλύψουμε και τα παλιά. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες φυσικά θα αναλυφθούν υπό το φως και με τους περιορισμούς των οικονομικών μας προβλημάτων. Και όπως είπα κατά την έναρξη της συζήτησης, Υπάρχει μεγάλη χρήση, μεγάλος αριθμός ενδιαφερομένων, γι' αυτό και περιμένω με ανυπομονησία τις τροπολογίες σας και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Δεν θα πρέπει όμως να λησμονούμε ότι στα θέματα της ενεργειακής απόδοσης υπάρχει μεγάλο περιθώριο καινοτομία για τις επιχειρήσεις μας και πολλές νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις θα πρέπει τα ευρωπαϊκά προϊόντα να αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία και φυσικά να δημιουργήσουμε και περισσότερες θέσεις εργασίας. Είναι μεγάλη ευκαιρία που μας προκύπτει. Γιατί ο καλύτερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εξοικονομήσουμε χρήματα είναι η ενεργειακή απόδοση. Ακούσαμε κάποια σχόλια και για τη χρηματοδότηση. Για την αφιέρωση περισσότερο κονδυλίων ε, και περισσότερο χρημάτων προκειμένου να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Όπως σας είπα, πολλά είναι τα σχόλια και πολλοί εμπλεκόμενοι. Ελπίζω μέσα από τις διαβουλεύσεις να συνεννοηθούμε, να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε μια στεναρή έκθεση που θα ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι. 5 Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία και η κατάθεση τροπολογιών και περνάω λοιπόν στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης το 15 βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης ε, εισηγητής ο συνάδελφο Λάνι, που του δίνει και κατευθείαν το λόγο για να ξεκινήσουμε το, τη συζήτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε, συνάδελφοι. Όντω. Όπως λέει και ο τίτλος, η βιομηχανική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι το θέμα μας. Κοιτάμε πώς δρούν οι φορείς ανταγωνισμού σήμερα. Είναι επιτακτικό καθήκον λοιπόν να ασχοληθούμε με τη βιομηχανική πολιτική. Να σας θυμίσω ότι τα ΙΠΑ επενδύουν δισεκατομμύρια, ότι ακόμα και η Κίνα ενισχύει την καινοτομία στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Και η Κίνα ασκεί έντονα επεκτατική πολιτική πρωτονηλών και η συνάντηση στην Ιαπωνία τόνισε και αυτή τη βιομηχανική πολιτική. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα στοιχεία αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι δεν μπορούμε πλέον να καθυστερούμε και να επιτρέπουμε στον εαυτό μας να συνεχίσουμε τη μη αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική των τελευταίων χρόνων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει άμεσα πάρα αυτά να ενισχύσουμε τη βιομηχανική βάση μας. Και επιπλέον υπάρχει και η πρόκληση της παγκόσμιας ε, κρίσης του κλίματος. Θα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτήν. Θα πρέπει με καλύτερο τρόπο να αξιοποιούμε τις πρώτες ύλες μας και τα δύο αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη νέα βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη. Τα τελευταία, τις τελευταίες εβδομάδες συνομίλησα με πάρα πολλούς συναδέλφους και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα σεμινάριο που διοργάνωσε η ομάδα μας. Ακούσαμε πολλές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και πολλές από αυτές τις συμπεριέλαβα στο σχέδιο έκθεσης. Είναι σαφές, συνάδελφοι, ότι αν θέλουμε να δράξουμε αυτή την ευκαιρία για τη βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη, θα πρέπει να είναι μια ενοποιημένη πολιτική σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση και την ε, ενοποίηση στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή είναι πολύ κατακαιρματισμένος ε, η κατακαιρματισμένη η κατάρτιση πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι ενοποιημένη η προσέγγιση. Και γι' αυτό λοιπόν προτείνω να δημιουργηθεί task force ομάδα κρούσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και συντονισμό, αρμόνιση μεταξύ των όσων πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Γιατί κατά τη διάρκεια της κρίσης φάνηκε ότι η εθνική πολιτική πολλές φορές παίρνει άλλη κατεύθυνση από την ευρωπαϊκή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, για να υπάρχει τέτοιος συντονισμός. Με τα δύο αυτά στοιχεία πιστεύω ότι θα πετύχουμε πολλά. Κοιτώντας λοιπόν τώρα συνάδελφοι τι πρέπει να γίνει. Προτείνω να επικεντρωθούμε σε μια οριζόντια δράση, στην οποία θα προσθεθούν ε, τομεακά, τομεακές και περιφερειακές πτυχές. Δεν θέλουμε επεμβατική πολιτική. Δεν είναι καλύτερη πολιτική αυτή από την πολιτική των επιχειρήσεων, αλλά Αφετέρου, η εμπειρία μας δείχνει ότι οι αγορές ρυθμίζονται μόνο τους με τον καλύτερο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια οριζόντια πολιτική. Και στο σχέδιο έκθεσης προσπάθησα να επικεντρωθώ σε τρεις βασικές ομάδες. Καταρχάς, καινοτομία και πολιτική για την καινοτομία. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο πολύ τη μεταφορά τεχνολογίας και τον τομέα των υλικών για να ενισχύσουμε πιο πολύ την καινοτομία. Και θέλουμε σύνδεση μεταξύ, για παράδειγμα, της προσέγγισης της ψηφιακής Ευρώπης και της παραδοσιακής προσέγγισης, προκειμένου όλες οι κατευθύνσεις τελικά να συμβάλλουν προς την ε, ανάπτυξη της καινοτομίας. Θα πρέπει να δοθούν πόροι τελικά προκειμένου να προωθηθούν ακόμα και καινοτομίε με υψηλό ποσοστό κινδύνου. Δεύτερη μεγάλη ομάδα, οι πόροι για την βιομηχανική δράση. Καταρχάς θέλουμε υλικού πόρους. Ασφαλώς. Και εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες. προσπαθούμε με διεθνείς συμβάσεις να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αρκετές πρώτες ύλες. Αλλά πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πόροι που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα χρειαστεί λοιπόν ένα γεωλογικό σύστημα γεωλογικής ανάλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξέρουμε τι πόρους διαθέτουμε. Θα πρέπει να αποτρέψουμε την εξαγωγή πολύτιμων πρώτων υλών με νόμιμο ή μη τρόπο. Και το τίθεται και το θέμα του ποιος διαχειρίζεται τις πρώτες ύλες. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, γιατί ε, προέκυψε, προέκυψε μια συγκεκριμένη δομή Έχουμε κάποια ολιγοπόλια τα οποία ασκούν έντονη πίεση στην βιομηχανική ανάπτυξη. Να δούμε λοιπόν τις πρώτες ύλες, τους πόρους, αλλά και την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων. Και αυτό αποτελεί βασικό θέμα για να είμαστε οικολογικά υπεύθυνοι και αποτελεσματικοί. Η νομοθεσία αποτελεί ένα εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε καλύτερα. Τρίτη μεγάλη, τρίτος μεγάλος ε, πόρος είναι το θέμα της εξειδίκευσης των εργαζομένων. Σήμερα σε κάποιες τομείς παρουσιάζεται το εξής πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να βρει κανείς εξειδικευμένους ε, εργάτες, εργαζόμενους. Και πάντα σκεφτόμασταν μήπως χρειάζεται εισαγωγή των εξειδικευμένων αυτών ατόμων. Χρειαζόμαστε λοιπόν σωστή εκπαίδευση, κατάρτιση, εξειδίκευση των ε, εργαζομένων στην Ευρώπη. Και εδώ πέρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πιο πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τρίτη ομάδα σε ό,τι αφορά την βιομηχανική κουλτούρα το βιομηχανικό πολιτισμό. Δεν έχουμε διαμορφώσει απαραίτητα την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τώρα όπως θα έπρεπε. Και αυτό από τι εξαρτάται. Για παράδειγμα, ότι πρέπει να βρούμε πιο καλά και να εντοπίσουμε με πιο καλό τρόπο τις ηγετικέ αγορές. Για παράδειγμα, στον ε, τομέα των δημοσίων συμβάσεων να τις ε, ανισχύσουμε. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να δοθεί όθηση σε καινοτόμα προϊόντα. Προϊόντα τα οποία υποστηρίζουν και τον ανταγωνισμό μας, αλλά και την περιβαλλοντική διάσταση. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τα προϊόντα αυτά. Αλλά και θέματα αναδιάρθρωσης θα πρέπει να μας απασχολήσουν πιο πολύ από ό,τι ως τώρα. Και μάλιστα εκ των προτέρων, προληπτικά να γίνει διάρθρωση όχι όταν θα έχει παρουσιαστεί πρόβλημα, για να δοθούν νέες πρόπτικες στις επιχειρήσεις. Στον τομέα λοιπόν αυτό χρειάζεται μια νέα κουλτούρα, νοτροπία ως προς την βιομηχανία και εδώ νομίζω ότι έρχεται και το θέμα των κρατικών ενισχύσεων πιστεύω ότι χρειάζεται διαφάνεια στις ε, κρατικές ενισχύσεις και χρειάζονται κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση καινοτόμων τομέων της βιομηχανίας προκειμένου να καταστούν και ανταγωνιστικοί αυτοί οι τομείς. Αυτό ασφαλώς δεν μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το εργαλείο αυτό. Πέρα από την ευρωπαϊκή διάσταση υπάρχει και η περιφερειακή διάσταση. Όλες οι μελέτες καταδεικνύουν ότι οι αποφάσεις για τις επενδύσεις της βιομηχανίας εξαρτώνται ιδιαίτερα από την ε, περιφερειακή διάσταση, δηλαδή από το πώς σχηματίζονται τα καινοτόμα δίκτυα, προκειμένου να σχηματιστούν περιφερειακά κλάστερ. Θα ήθελα λοιπόν να ενισχύσουμε αυτές τις περιφερειακές ε, ομάδες τα περιφερειακά κλάστερ προκειμένου να τονώσουμε και την βιομηχανία σε αυτό το επίπεδο. Πέρα από την οριζόντια προσέγγιση, θα ήθελα και στους μεμονωμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για τη βιομηχανία να αναλυφθούν τομεακές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, προκειμένου να προωθηθεί η καινοτομία αλλά και κινητικότητα, αλλά και σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες ε, έχουν καταστεί πολύ σημαντικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις αναφορικά με την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων και η Κίνα επενδύει πάρα πολλά στον κλάδο αυτόν. Και δεν είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτό συμβαίνει υπό δίκαιους, σωστούς, θεμητούς όρους. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ακολουθήσουμε και μια τομεακή προσέγγιση. Και είμαι αισιόδοξο ότι όλοι από κοινού θα μπορέσουμε να δημορφώσουμε μια νέα φρέσκια, αν θέλετε, βιομηχανική πολιτική, προκειμένου να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι τις προτάσεις αυτές θα μπορέσουμε να τις ενσωματώσουμε και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα δημοσιευθεί στις 13 ε, Οκτωβρίου προκειμένου να προκύψει ένα κοινό κείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Λέει ο Πρόεδρος, ο συνάδελφος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Λάγκε, ο οποίος μας υπέβαλε και ένα πρώτο σχέδιο εργασίας και σε σχέση με το πρώτο αυτό έγγραφο η έκθεση είναι πολύ λιγότερο παρεμβατική και πολύ πιο ισορροπημένη. Ξέρω, βλέπω μάλλον ότι το θέμα των πρώτων υλών ε, το τονίσατε πιο καλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τομεακή προσέγγιση. Πρέπει να πω ότι βελτιώθηκε πολύ το έγγραφο και χαίρομαι που προσπαθείτε να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ έρευνας και καινοτομία και ανταγωνιστικότητας αφετέρου. Ζητάτε τον ορισμό της καινοτομίας, έναν ευρύ ορισμό της καινοτομίας. Εγώ θα πρότεινα η καινοτομία να περιλαμβάνει όλα όσα α, συνεπάγεται η αξιοποίηση χρηματική μιας ιδέας. Από τη γνώση δηλαδή βγάζουμε χρήματα υπό τη μορφή μιας υπηρεσίας ενός προϊόντος. Επί της αρχής θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα δημορφωθούν τα κίνητρα για την ε, καινοτομία. Υπάρχουν πολλά προγράμματα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι απλά τα πράγματα. Για παράδειγμα, η ηλεκτρική κινητικότητα μπορεί να προωθηθεί τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να προωθηθούν με την ε, δωρεάν στάθμευση των αυτοκίνητων αυτών. Μιλάμε για προγράμματα, για σχέδια τα οποία μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμο μεγάλο αντίκτυπο. Αυτό που κάπως λείπει θεωρώ είναι η αναφορά στις αγορές. Δηλαδή το από πού προέρχεται ένα προϊόν. Νομίζω ότι στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανικής πολιτικής θα πρέπει να εξετάσουμε το ποσοστό της παραγωγής που προέρχεται από την ε, Ένωση. Και αυτό γίνεται με την επισήμανση, με το labeling. Οι Γάλλοι, οι Ιταλοί είναι υπέρ της λύσης αυτής, οι σκανδιναβικές χώρες είναι κατά. Να το συζητήσουμε, αλλά αυτό δημιουργεί, δημιουργεί διαφάνεια για τον ε, καταναλωτή. Ξέρει από πού προέρχεται το προϊόν που αγοράζει. Επίσης, Αναφέρεστε συχνά στην Κίνα. Γι' αυτό και εγώ θα ταχθώ υπέρ μιας εταιρική σχέσης ε, με την Κίνα. Ας μην ε, κλείνουμε τα μάτια. Ως ε, Ευρώπη θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Κίνα. Αυτό είναι καλό, ωφέλιμο, αλλά και παράλληλα επικίνδυνο. Είναι καλό επειδή έτσι καταφέραμε να χρησιμοποιήσουμε και εμείς να αξιοποιήσουμε εμείς ως Ευρώπη την ε, άνοδο της Κίνας, αλλά είναι επικίνδυνο γιατί οι Κινέζοι θα απαιτήσουν σε αντάλλαγμα μεταφορά της γνώσης μας προς την Κίνα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει και ένα θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, οι Κινέζοι τις ε, γερμανικές ευρεσιτεχνίες. Τις χρησιμοποιούν όμως επιθετικά και κατά τη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια σχετική συμφωνία. Ίσως θα μπορούσε να προκύψει ένα κοινό δικαστήριο. Αυτό που είναι καθοριστικό ωστόσο είναι να είναι εταίρος μας εκείνα. Σε θέματα εκπαίδευση, για παράδειγμα, ίσως κάποια στιγμή να δημιουργηθεί και μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου. Αλλά είναι πολύ βασικό το στοιχείο αυτό για την βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης. Κάτι άλλο που σχετίζεται και με την Κίνα αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο πόλεμος του ταλέντου. Δηλαδή, πώς ε, θα μπορέσουμε στην Ευρώπη να αντιμετωπίσουμε την δημογραφική τάση που δημιουργεί ελλείψεις σε εξειδικευμένο ε, προσωπικό. Μηχανικούς. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, αναφέρεται σε μελέτες ότι θα λείψουν στο μέλλον 95.000 ε, μηχανικοί. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και δεν θα καταφέρουμε σε βιομηχανικό επίπεδο να επιβιώσουμε αν δεν συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη. Δεν μπορούμε να μην αγωνιστούμε. Θα πρέπει να υπάρξει να γίνουν έντονες προσπάθειες. Γιατί η Ευρώπη ζει από την τεχνολογία, αλλά ζει και από την ε, στάση που επιδεικνύει προς τους ξένους. Άρα θα πρέπει να δείξουμε, ε, καθήκον μας είναι να το διαβιβάσουμε αυτό προς τους ε, πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος, η κυρία Κρουστέτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε ως και για την εκμέρους του ΕΛΚ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Λάγκε. Να τον ε, συγχαρώ για την έκθεσή του και να πω ότι σε ορισμένα σημεία θα μπορούσαμε να είμαστε πιο διεξοδικοί. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Λάγκε μας μίλησε για το πρόβλημα των κρατικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις. Όντως είναι μια δυσκολία που αντιμετωπίζουμε γιατί ισχύουν ευρωπαϊκοί κανόνες που δεν είναι όμως διεθνείς κανόνες και έχουμε, αντιμετωπίζουμε στρέβλωση ανταγωνισμού, μερικές φορές κατάσταση επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αυτό το θέμα των κρατικών ενισχύσεων και να τις εξετάσουμε υπό το πρίσμα της ανάγκης διατήρησης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Θέλουμε Ευρωπαίους πρωταθλητές ε, της βιομηχανίας μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Airbus θεωρείται ως επιτυχημένη επιχείρηση και είμαστε όλοι περήφανοι για αυτή. Και σήμερα δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια επιχείρηση εξαιτία των πολύ αυστηρών ε, ισχυών των κανόνων ανταγωνισμού. Και εκεί έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα πρέπει να το επιλύσουμε. Είναι ανησυχητικό. Αν δεν μπορούμε πια να δημιουργήσουμε νέους ευρωπαίους πρωταθλητέ, τότε ε, τι καταφέραμε. Επίσης υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότησης. Ο εισηγητής φυσικά μίλησε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά υπάρχει και το θέμα των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Η βιομηχανία χρειάζεται μια μακρο, μακροπρόθεσμη, μακρόπνοη πρόπτικη, γιατί η βιομηχανία απεχθάνεται την αβεβαιότητα δεν αντέχει την ανασφάλεια. Και αυτή την αβεβαιότητα διαονίζουμε μέσω της νομοθεσίας μας, ακόμη και στα πλαίσια της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχεια με το μείον 20, μείον 30 έφερε σε απελπισία τους επιχειρηματίες γιατί δεν ξέρουν πώς θα προβλέψουν το μέλλον και προς τα πού να στρέψουν τις επενδύσεις τους θα πρέπει όταν υιοθετούμε μία στάση να την κρατούμε με αποφασιστικότητα και να μην αλλάζουμε κάθε τρει και λίγο. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό και την απασποσβατοποίηση της αγοράς με, την... Ε, με προδιαγραφές και να διαφυλάξουμε και τα εργοστάσια μας. Πώς νοείται βιομηχανική πολιτική χωρίς εργοστάσια. Γνωρίζουμε όλοι το πρόγραμμα Γαλιλαίο έχουμε 14 από τους 30 δορυφόρους που με διαγωνισμό δόθηκαν σε μια γερμανική μικρομεσαία επιχείρηση. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η μικρομεσαία επιχείρηση έδωσε υπεργολαβία στις Ηνωμένε Πολιτείες 14 από αυτούς τους δορυφόρους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιο είδους ανάθεση και διαφυγή. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερη ενημέρωση ε, για την ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων και αυτό είναι το βασικό θέμα του Made in Europe. Θα πρέπει να προαγάγουμε την ποιότητα της βιομηχανίας μας. Σε ό,τι αφορά το διοικητικό άκθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, το συζητάμε χρόνια ολόκληρα, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα. Επίσης, μιλήσαμε για τις συμπράξεις κρατικού και ιδιωτικού κεφαλαίου. Έχουμε και την έκθεση Καρβάλιο για την απλούστευση και την εφαρμογή του ερευνητικού προγράμματος πλαισίου. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολύ απτά. Είπαμε ότι η καινοτομία θα επιτύχει μόνο χάρη στη σωστή κατάρτιση και επιμόρφωση. Όπως είπαμε, στην αεροναυπηγική χρειαζόμαστε 12.000 μηχανικούς το χρόνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 9.000 ε, μηχανικούς αεροναυπηγικής το χρόνο. Υπάρχει έλλειμμα στην περίπτωση αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε νέους κλάδους στις, στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Και το θέμα της ε, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας είναι σημαντικό. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρυστεχνίας που το περιμένουμε χρόνια ολόκληρα, αλλά εξαιτία μεταφράσεων το θέμα έχει καθυστερήσει. Φυσικά τα διπλώματα ευρεσιτεχνία δεν πρόκειται να προστατεύσουν τα πάντα. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Σε ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκή Ένωση ανακαλύψαμε κινέζικα ελαστικά που ε, διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά και μιμούνται κάλλιστα τα ευρωπαϊκά ελαστικά, καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνία, αλλά είναι πολύ κατώτερη ποιότητα από τα ευρωπαϊκά ελαστικά και είναι και επικίνδυνα. Θα πρέπει δηλαδή να, ενισχύσουμε του ελέγχου Σήμερα η έλεγχοι στα σύνορα είναι ελλειπείς. Μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά ε, ψευδεπίγραφα φάρμακα ή παραποιημένα προϊόντα. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να τα αναχαιτήσουμε. Και υπάρχει και το θέμα της εξωτερικής διάστασης της βιομηχανικής πολιτικής. Νομίζω ότι αξίζει ολόκληρο δικό της κεφάλαιο με το θέμα της πρόσβασης της αγοράς. Και χθε μιλήσαμε και για την αρχή τη αμοιβαιότητα. Θα πρέπει να ισχύει η αρχή τη αμοιβαιότητα για να αποφευχθεί το κοινωνικό ή το περιβαλλοντικό dumping. Θα ήθελα, εν κατακλείδη, να αναφερθώ στο θέμα της ε, ετικετοθεσίας των προϊόντων και της ανάγκης ε, σωστής σήμασης, της καταπολέμησης επίσης της παραποίησης. Έχουμε την ε, πολύ καλή έκθεση Μουσκαρντίνη στην Επιτροπή Εσωτερικού Εμπορίου. Καλό θα ήταν να εμπνευστούμε και από αυτή την έκθεση. Ο εισηγητή αναφέρθηκε και στο θέμα των πρώτων υλών. Όντω έχουμε ένα κατάλογο με 14 πρώτε ύλε, ένα κατάλογο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατανάλωσή του προβλέπεται να τριπλασιαστεί την επόμενη 20 ετία και χάρη στη χρήση περιβαλλοντικής ε, πολιτικής. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πραγματική εξωτερική πολιτική βιομηχανική για να προστατεύσουμε τους φυσικούς μας πόρους και τις πρώτες μας ύλες. Ο εισηγητής μίλησε για την οριζόντια προσέγγιση αλλά και για την ανάγκη κλαδικής προσέγγισης. Χρειαζόμαστε και τις δύο προσεγγίσεις, και την ε, οριζόντια και την τομεακή. Θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες για να εμπλουτίσω την έκθεση, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να προτείνουμε στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία γνήσια στρατηγική, όχι βιομηχανική πολιτική, μία βιομηχανική στρατηγική, γιατί αυτό πραγματικά χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Κοσνόφσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, είμαι πεπισμένος ότι η όλη συζήτηση η θεωρητική για τη βιομηχανική πολιτική μας ε, ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης είναι πάρα πολύ ευρεία. Είναι δύσκολο να επικεντρωθούμε στην ουσία του θέματος. Πρέπει να αποφύγουμε τις θεωρητικές, τα θεωρητικά αποφθέγματα και να μην καταλήγουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κάποια σχόλια τώρα για τους τομείς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την βιομηχανική μας, τις βιομηχανικές μας δυνατότητες για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Για την έρευνα επίσης. Η έρευνα μπορεί να βοηθήσει την βιομηχανία εκεί όπου τα δημόσια κονδύλια δεν επαρκούν. Είναι δύσκολο να εξεύρουμε την σωστή χρηματοδότηση, να στηρίξουμε την βιομηχανία, η οποία ούτως ή άλλως λειτουργεί σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε έναν βιομηχανικό τομέα μόνον και να στηρίξουμε αυτόν. Όπως είπαν κι άλλοι συνάδελφοι, είναι σημαντικό το πόσο μπορούν να βοηθήσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συγκεκριμένα για την επαγγελματική κατάρτιση, την ε, εκπαίδευση των δυναμικού. Εδώ υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και μπορούμε να βοηθήσουμε τον ε, σχολικό τομέα, τον τομέα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε με τις επόμενες γενιές να είμαστε έτοιμοι Πρέπει όμως από τώρα να προλάβουμε. Ξέρουμε ότι ένας αεροναυπηγός ή ένας ερευνητής στον τομέα της ενέργειας ή ένας μηχανικός που ασχολείται στις, ε, με τις εφαρμογές της αεροδιαστημικές δεν μπορεί να εκπαιδευτεί σε τρία χρόνια. Χρειάζεται τουλάχιστον μια πενταετία ε, μαθημάτων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι και να έχουμε άτομα με δεξιότητες που θα μπορούν να μας βοηθήσουν τα καινοτόμα βήματά μας να τα υλοποιήσουμε. Δεν είναι απλό κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη όμω δεν μπορεί να κοιτάζει μόνο τα ποσοστά, τι ποσότητε, του αριθμού των πτυχιούχων και διπλωματούχων. Πρέπει να μα απασχολούν και πραγματικέ δεξιότητε και ικανότητε των ατόμων να εργάζονται σε αυτό τον τομέα, να προχωρούν και να προοδεύουν. Πρέπει λοιπόν έτσι να βοηθήσουμε τη βιομηχανία ώστε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη. Το σκηνικό βεβαίω τη παγκοσμιοποιημένη αγορά ναι, χρειαζόμαστε φιλόδοξους στόχους, αλλά σίγουρα με την επιτυχία των προϊόντων μας, με δεξιότητες, με νέα σύγχρονα προϊόντα ελκυστικά, τότε θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Σε αυτή λοιπόν την έκθεση ίσως λείπει ένα στοιχείο. Δηλαδή, κάποια περισσότερα σχόλια ή έστω μια απορία για το κατά πόσον εμείς ως θεσμικά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν θα επιβαρύνουμε διοικητικά την βιομηχανία. Μην περιπλέξουμε περαιτέρω τη ζωή τους. Να μην δημιουργήσουμε εμείς φραγμούς. Να μην επιβάλλουμε άχθος περιττό όπως ε, με τα ζητήματα της ετικετοθεσίας. Εδώ μιλάμε για επιπλέον κόστο που κάποιε φορέ θα πρέπει να καλύψει η βιομηχανία. Άρα από οικονομική άποψη ένα 10% κάθε επιμέρου προϊόντο θα πρέπει να κατευθύνεται στην κάλυψη του διοικητικού κόστου, Εφόσον εμεί προβλέψουμε τέτοιες διοικητικέ υποχρεώσει. Εάν λοιπόν κοιτάξουμε τι προκλήσει του μέλλοντος, που θα πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση επιφυλακτικοί, να είμαστε συνετοί. Ιδάλλως θα πληγεί η ανταγωνιστικότητά μας. Μπορεί να υποβαθμιστεί αυτή η ανταγωνιστικότητα. Και να μην πολλούνται αρκετά τα προϊόντα μας στην παγκοσπημένη αγορά. Για ένα παράδειγμα τώρα που ήθελα να αναφέρω από την Δημοκρατία της Τσεχίας. Μιλάμε για στήριξη, για την στήριξη των οικολογικών εφαρμογών, των πράσινων τεχνολογιών. Στην Δημοκρατία της Τσεχίας έχουμε μια πολύ καλή εμπειρία από όλα αυτά, διότι η στήριξη για τα φωτοβολταϊκά δεν ε, έχει οργανωθεί αρκετά καλά και ήδη του χρόνου θα έχουμε ένα 20% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τέτοιες πηγές. Η κατεύθυνσή μας λοιπόν είναι σωστή, αλλά τελικά δεν καταλήξαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Φοβόμαστε ότι μπορεί να πληγεί η βιομηχανία μας, η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας στο διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει εξέταση αυτού του θέματος, το πώς επηρεάζεται, πώς επηρεάζει η παγκοσμιοποίηση δηλαδή και να προσπαθήσουμε εντατικά να καταλήξουμε σε ουσιαστικά αποτελέσματα στη μελλοντική επιτυχία της ευρωπαϊκής οικονομίας να εξασφαλιστεί. Μιλάμε για μια βιομηχανία κινητική που μπορεί να δώσει οικονομικά ωφέλη στην Ευρώπη. Ο τραπεζικός κλάδος είναι δευτερογενής. Όμως η δυνατότητα να εξελιχθούμε σε οικονομικό επίπεδο και να προχωρήσουμε στο προσκήνιο το οικονομικό είναι κάτι που πρέπει να το εξασφαλίσουμε ως δυνατότητα και στον βιομηχανικό μας κλάδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλές καλές παρατηρήσεις βρίσκω στο σχέδιο έκθεσης του συναδέλφου Λάνε. Και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την χρήσιμη δουλειά που έκανε. Και νομίζω ότι ιδιαίτερα στο επίπεδο των στόχων και των οραμάτων αναφορικά με την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια διαφωνίας. βρισκόμαστε σε μια φάση πράσινης εισαγωγικά πράσινου οράματος και μιλάω για πράσινο όραμα αναφορικά με την οικολογική διάσταση, όχι με την πολιτική. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί την απαραίτητη βάση προκειμένου στο μέλλον στην Ευρώπη να διαμορφώσουν μια βιώσιμη, βιώσιμη ε, βιομηχανική πολιτική και να μην υπάρξει μετακατάσταση σε άλλες περιοχές του κόσμου. Πέρα από αυτά τα οράματα όμω και από αυτή τη μελλοντική διάσταση, θα ήθελα να εστιαστώ στη βασική αντίληψη της βιομηχανικής πολιτικής, στο βασικό της ορισμό και να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Δεν είμαι υπέρ της, του παρεμβατισμού σε κρατικό επίπεδο, ούτε υπέρ του προστατευτισμού. Η κυρία Γκροστέτ έθιξε το θέμα μιας γερμανικής εταιρείας η οποία είπε ότι έφτασε μέχρι να πουλήσει τέτοια θέματα παραγωγής προς τους Αμερικανικούς, Αμερικανούς. Λίγο περίεργο μου φαίνεται αυτό. Είναι προβληματική αυτή η αντίληψη της βιομηχανικής πολιτικής, θεωρώ. Τι έχουμε δηλαδή με τους Αμερικανούς. Θα ήθελα λοιπόν να τονιστεί η οριζόντια προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να θέσουμε κάποιες πολιτικές αρχές. Χωρίς να επισερχόμαστε σε λεπτομέρειες απαραίτητα κάθε φορά. Και κατά τρίτον θεωρώ ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα των μέσων και των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Να δούμε ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι τομεί. Εγώ είμαι νυφάλιος. Δεν είναι δυνατόν να κάθομαστε και να γράφουμε τι πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση, γιατί δεν πρέπει να γίνει σε άλλες περιπτώσεις. Θα πρέπει να δούμε τι πραγματικά μπορεί να επιλέξει η Ευρώπη, ποια είναι η καλύτερη, μεγαλύτερη δύναμη της, Ευρω... Ευρώπης. Και όπου δεν έχουμε αρμοδιότητα, όπου δεν είμαστε οι πιο ικανοί, να αφήσουμε τους άλλους. Αυτά νομίζω ότι θα καθορίσουν μια αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βέιμπερ. Ευχαριστώ. Η έκθεση του συναδέλφου είναι ιδιαίτερα πλούσια και πολύ πυκνή. Θα την εμπλουτίσουμε περαιτέρω με τροπολογίες. Δεν θα περάσω τώρα σε λεπτομέρειες. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή όσα είπε ο συνάδελφος για την ανάγκη να έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική, βιομηχανική πολιτική ολοκληρωμένη και επίση άκουσα προσεκτικά αυτά που είπε για την ανάγκη να συμπεριληφθεί η συνιστόσα η κοινωνική και η περιβαλλοντική στι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών, τι εμπορικέ μα συμφωνίε. Είναι πολύ σημαντικό. Επίση, την προσοχή που δίνει στο θέμα των πόρων. Το θεωρώ και αυτό εξίσου σημαντικό και θα πρέπει να μας απασχολήσει στις συζητήσεις μας. Τώρα ήθελα και εγώ να σταθώ σε μερικές παρατηρήσεις. Πιστεύω ότι σε ορισμένε περιπτώσει θα μπορούσαμε να τι συμπληρώσουμε και με τροπολογίε. Ε, πρώτον, δεν νομίζω ότι σε μια τέτοια έκθεση για τη βιομηχανική πολιτική μπορούμε να αποφύγουμε το θέμα τη χρηματοδότηση. Δεν γίνεται. Πρόκειται για ένα κριτήριο αξιοπιστία μας. Τα χρήματα είναι ένα όπλο για τον πόλεμο ε, όπως έλεγε ένας ε, φιλόσοφος, νομίζω Μακιαβέλη, αλλά και για την πολιτική ισχύ αυτό και σίγουρα χρειάζεται για τη βιομηχανία. Μιλάμε εδώ για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με την προοπτική του 2013. Ε, από την πλευρά λοιπόν του ευρωπαϊκού προπολογισμού πρέπει να αναζητήσουμε πηγές χρηματοδότησης. Τώρα συμβαίνει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μπαρόζο, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης να μιλά υπέρ των πηγών που έχουν δυνατότητες αναγνωρισμένες για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ε, ευρωομόλογα και μπορούν να δώσουν χρηματοδότηση για μεγάλα έργα υποδομών. Έκανε επίσης ε, ε, κάποιους πενιγμούς για φορολογίες ε, κάποιων ε, συναλλαγών. Και εδώ δεν μιλάμε για μια προσέγγιση αριστερίστικη, μιλάμε για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πράγματι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυνατότητα χρέωσης και εάν συμφωνήσουμε με αυτά που μας προτείνονται στην έκθεση αυτή του κ. Λάγκε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι θα αντιμετωπιστεί και το ζήτημα τη χρηματοδότηση. Ιδάλω θα καταλήξουμε στα δύο αποτελέσματα όπω με τη στατιακή του Λισαβόνα, Μια σειρά από ευγενεί προθέσει που παρέμειναν όμω νεκρό γράμμα, ε, στο κείμενο, στα χαρτιά δηλαδή. Και ανατέθηκαν στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη ξέρετε ότι έχουν επιδοθεί όμω σε καλυστία μεταξύ τους, ένα διαγωνισμό ομορφιά για ε, να δουν ε, ποιος θα πάρει τα μεγαλύτερα ποσά από τον προπολογισμό. Εδώ λοιπόν ε, υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνε και δεν μπορούμε να έχουμε και αυταπάτες για το θέμα της χρηματοδότησης. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μιλάμε για τον εύρο, το, τη μοντελική στήλη όλων αυτών και το κλειδί της αλήθειας στην ουσία. Πρέπει να τα πάρουμε όλα αυτά πολύ σοβαρά. Εάν θεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι τελείως διαφορετικό, άσχετο, ότι δεν αποτελεί μέρος των ανησυχιών της Επιτροπής μας και δεν αντικατοπτριστεί στη συγκεκριμένη έκθεση, θα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα σίγουρα, αλλά στη φάση της υλοποίησης δεν θα έχουμε σοβαρή επιτυχία. Μια δεύτερη παρατήρηση τώρα. Και εδώ έχουμε ένα από τα θετικά στοιχεία της έκθεσης ό,τι αφορά τον συντονισμό, τη συνεργασία των βιομηχανικών πολιτικών των κρατών μελών, και σε αυτό που ονόμασε ο εισηγητής μας ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Πρέπει να αποφύγουμε τις επαναλήψεις στην Ευρώπη, τις επικαλύψεις προσπαθειών. Δηλαδή, εάν η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία συνεργαστούν για να συλλάβουν, να σχεδιάσουν και να παράγουν ένα αυτοκίνητο οικολογικά καθαρό, υβριδικό και πράσινο, ε, θα πρέπει να το κάνουν αυτό, να τους επιτραπεί, να κάνουμε τα ίδια που κάναμε στην αεροναυπηγική, στο διάστημα και σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή να συνεργαστούμε, να την προωθήσουμε τη συνεργασία. Όταν δεν υπάρχουν πολλά μέσα, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην διασπείρονται δεξιά και αριστερά, αλλά να συνενώνονται μια τρίτη τώρα παρατήρηση και είναι και αυτό ένα σημείο που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Η επιτυχία της βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρώπη θα εξαρτηθεί και από την νομισματική μας πολιτική αρκεί να είναι εύστοχη. Και επίσης και από την πολιτική ανταγωνισμού που θα πρέπει να είναι λιγότερο δογματική από αυτή που ακολουθεί για την ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νομισματική πολιτική για να είναι εύστοχη προφανώς θα πρέπει να μην στραφεί προς ένα υπερτιμημένο ευρώ που αντιμετωπίζει ένα γεν υποτιμημένο και ένα δολάριο που και αυτό μπορεί να υποτιμηθεί μακροπρόθεσμα, διότι όλες μας οι προσπάθειες θα καταστραφούν σε αυτή την περίπτωση από, την, ε, από τον αθέμητο νομισματικό ανταγωνισμό. Πρέπει λοιπόν, απαραίτητο κατά την άποψή μου, όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία και η Κίνα ακολουθούν νομισματική πολιτική συνεπή, έχουν πολιτική συναλλαγών και ισοτιμία, θα πρέπει και εμεί αυτό να κάνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε ο μόνο οικονομικό παράγοντα στον κόσμο που να μην έχει τέτοια πολιτική. Παρομοίω, ε, όπω υπόθηκε προηγουμένω, αλλά το επαναλαμβάνω κι εγώ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εφόσον αποφασίσουμε ότι η βιομηχανική μας πολιτική είναι προτεραιότητά μας, θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή την απόφαση. Διότι πραγματικά είναι πολύ ωραία να τα γράφονται αυτά στα κείμενα, όμως πρέπει να, να, ξέρουμε ότι η βιομηχανική βάση της Ευρώπης απειλείται, χάνουμε μερίδια από την αγορά. Ε, ε, στον τομέα της βιομηχανίας, με μόνη εξαίρεση τη Γερμανία που όμως είναι εξαίρεση για την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν ε, η επαναβιομηχανοποίηση να γίνει προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η συμμετοχή όλων ε, στην βιομηχανική προσπάθεια για να προκύψουν εθνικοί πρωταθλητές είναι μια προσπάθεια που πρέπει να στηριχθεί. Η Επιτροπή καταδικάστηκε τρει διότι ε, ε, απαγόρευσε συγχωνεύσεις ενώσει ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δεν θα σας απαριθμίσω τώρα τις περιπτώσεις, όμως έτσι δεν θα επιβεβαιώσουμε την ανάδυση Ευρωπαίων πρωταθλητών που θα μπορούσαν να γίνουν και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Διότι ένα διεθνή πρωταγωνιστής πρέπει πρώτα να είναι πρωταγωνιστή και στην δική μα την Ήπειρο, την Ευρώπη, για να πετύχει έξω. Ε, αυτά για τις πτυχές του του ανταγωνισμού. Τώρα στην, ε, στην εισήγηση του ο κύριος Λάγκε μίλησε και για το τι συμβαίνει με τις πράσινες, τις οικολογικές ε, τεχνολογίες. Πράγματι η Κίνα αποφάσισε να είναι ο πρώτος παγκόσμιος παραγωγός σε αυτόν τον τομέα. Όπως και σε όλους τους άλλους, έτσι, γιατί οι Κινέζοι έχουν ε, δεν ασχολούνται με τους διάβλους, τις εξειδικεύσεις και τις ε, ειδικότητε, τις λεπτομέρειες. Θέλουν να είναι πρώτοι και θα το πετύχουν. Έχουν ένα μαζικό πρόγραμμα, ένα πολύ ογκώδες πρόγραμμα επενδύσεων, 580 δις δολάρια και τα 38% αυτού του χαρτοφυλακίου προορίζονται για τις ε, τεχνολογίες του μέλλοντος και ειδικά τις πράσινες. Οι πράσινες λοιπόν τεχνολογίες θα είναι θέματα όλων των μορφών του dumping χωρίς καμία εξαίρεση, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού. Ε, οι κεντρικές τράπεζες δηλαδή, οι κρατικές, δίνουν στις κρατικές ε, εταιρείε, όλα τα απαραίτητα δάνεια με μηδονικό επιτόκιο, επιστρέφονται τα δάνεια αυτά και προφανώ γι' αυτό οι Κινέζοι ήρθαν πρώτοι στην παραγωγή ε, ενέργεια από βολταϊκέ πηγέ, ε, την παραγωγή αιωλική ενέργεια και κατακλείζουν την αγορά με τα προϊόντα του. Η ερώτησή μου λοιπόν προ τον εισηγητή είναι εμεί τι κάνουμε υπό αυτέ τι συνθήκε. Εδώ μιλάμε για τις βιομηχανίες του μέλλοντος που με μεγάλα ποσά επενδύονται. Εμείς ε, θα πάμε στον ΠΟΕ, θα ζητήσουμε μια ρήτρα διασφάλισης ε, κατά των επιδοτήσεων, του ντάμπινγκ. Στην έκθεση πρέπει κάτι να λέγεται, σαφώς. Εγώ δεν είμαι υπέρ του προστατευτισμού. Είμαι τελείω εχθρικό. Όμω θέλω να, αυτο... να προστατεύσουμε του εαυτού μα όπω κάνουν και άλλοι. Οι Αμερικανοί ξέρουν να προστατεύουν του εαυτού του που είναι τόσο φιλελεύθεροι. Και οι, οι Ιάπωνε το ίδιο. Ε, δεν θα μιλήσω για του Κινέζου που δεν δίνουν διάρα για του υπόλοιπου, αλλά είναι υπερπροστατευτικοί με τον εαυτό του. Ε, πρέπει λοιπόν να ξέρουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μα. Δεν το κάνουμε για την ώρα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε υποδειγματικοί ώστε όλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά μα σε έναν άκρατο φιλελευθερισμό. Μα είναι φιλελέ εκ μέρου μα. Ο καπιταλισμό αναπτύσσεται στην Κίνα και δεν είναι φιλελεύθερο καπιταλισμό. Είναι αφέλη να το πιστεύουμε αυτό. Είναι καπιταλισμό κρατικό. Βασίζεται σε γίγαντε κρατικού και διαθέτει τεράστια κεφάλαια τα οποία συνδέονται με την αδυναμία τη ε, κατανάλωση, με την ε, περιορισμένη κατανάλωση. 35% είναι η κινέζικη κατανάλωση του δικού του ΑΕΠ. Ενώ σε εμά έχουμε 60, 55% στι ΗΠΑ 60%. Έχουμε λοιπόν εδώ δύναμη και έχουμε δικαίωμα να αλλάξουμε το δικαίωμα, το, τους κανόνες μας για, τους, ε, για τις κρατικές προμήθειες. Τους διαγωνισμούς. Εάν δεν αλλάξουν οι σχετικοί κανόνες δεν θα πετύχουμε αυτά που νομίζουμε. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει τον λόγο. Μετά έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή. Δηλαδή ενάμιση λεπτό για τον καθένα. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα πρέπει να συντομεύσουν ο συνάδελφο Μπρέντ. Ή συνάδελφος Μπρέντ. Φαν Μπρέντ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ε, ελπίζω καλά να σα κατάλαβα, γιατί προσπαθώ να καταλάβω τα γερμανικά σα. Είπατε να είμαι σύντομη. Πολλά ακούσαμε ήδη, που με βρίσκουν σύμφωνοι. Να συγχαρώ όμω τον ε, εισηγητή για την πολύ ισορροπημένη έκθεση. Αν κάπου πρέπει να εφαρμόσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη, είναι στην ε, βιομηχανική πολιτική και νομίζω ότι πολύ καλά τα πέτυχε αυτά ο εισηγητής. Να τονίσω ένα στοιχείο το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι θα είναι πολύ βασικό να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση που είναι απαραίτητη για τη βιομηχανία μας να μετατραπεί, να γίνει μια άλλη βιομηχανία. Πολλά χρήσιμα μας αναφέρει ο εισηγητής. Μιλάει για τις πρώτες ύλες και πόσο σημα... σημαντικές είναι. Δεν θα πρέπει να το παραμελούμε αυτό. Γιατί οι επιχειρήσεις μας διαρκώς αναζητούν τρόπους ε, εξοικονόμησης ε, και κυρίως εστιάζονται στα εργατικά, αλλά τα εργατικά είναι το 20% του συνολικού κόστους για τη βιομηχανία. Το 40% είναι οι πρώτες ύλες. Άρα, από όλες τις απόψεις θα πρέπει να κοιτάξουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και θα υποβάλω τροπολογίες που θα έχουν να κάνουν με τις πρώτες ύλες και θα πρέπει να φροντίσουμε για τις ε, πρώτες ύλες, γιατί δεν είναι απεριόριστες και δεν πρόκειται για θεωρητικές, θεωρητικά σχέδια. Πρόκειται για σχέδια τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν πρακτικά και τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε. Επόμενος ε, ομιλητής. Ο κύριος ε, Ενά. Δεν κατάλαβα το όνομά μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πολύ γρήγορα είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία που πήρε η συζήτηση. Και θα προσέξατε ότι υπάρχει μία ε, ρηξικέλευθη αλλαγή της γαλλικής θέσης και της Συμβίας. Όλοι διαπιστώσαμε ότι από την κρίση η Γερμανία τα κατάφερε καλύτερα από τη Γαλλία, γιατί επέλεξε ένα σημαντικό εθνικιστικό βιομηχανισμό, βιομηχανική πολιτική γιατί ε, πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, παράγει και καταναλώνει, σε αντίθεση με τη Γαλλία που εισάγει τα περισσότερα αυτοκίνητα. Έχουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις της Γερμανίας ε, και ως προς τη χρήση του προϋπολογισμού και ως προς την ε, εξυπηρέτηση των πολιτών. Θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί και η ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί λέμε η διαχείριση των αποβλήτων να γίνεται κοντά στην παραγωγή τους και δώσαμε επιδοτήσεις για να γίνεται διαχείριση αποβλήτων κοντά στην παραγωγή τους. Θα πρέπει και τα βιομηχανικά προϊόντα να παράγονται κοντά στο χώρο κατανάλωσής τους ώστε να αποφύγουμε τα λύκες ε, ή ε, δεξαμενόπλια να κυκλοφορούν ε, αντί να είναι κοντά στον τόπο κατανάλωσης. Επίσης, είπαν ορισμένοι προσοχή να αποφύγουμε τον παρεμβατισμό. Όπως είπαν όμω η κυρία Γκροστέτ και ο κύριος Βέμπερ είπε ας μην είμαστε αφελεί. γιατί αν πάμε όλο με το σταυρό στο χέρι θα καταφέρουμε τίποτα. Οι Αμερικανοί έχουν μαζικές ενισχύσει. και κάνουν ό,τι μπορούν για να κερδίσουν ε, Αγορέ, Για να μην πούμε για τις επιλογές. Οι ίδιες ε, επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, που βρίσκονται στην Κίνα κάνουν ό,τι μπορούν για να διεκδικήσουν ένα μερίδιο αγοράς. Ναι, στην ε, ευρωπαϊκή στρατηγική και όχι στο νόμο της αγοράς. Και θα πρέπει να επαναπατρίσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ευχαριστώ κυρία Χέρτσοκ. Ευχαριστώ. Κάθομαι στα αριστερά, δύσκολο να με δείτε κατευθείαν. Δύο ζητήματα πολύ σύντομα. Νομίζω είναι πολύ καλή κίνηση τελικώς ε, να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη την εσωτερική αγορά, την περιβαλλοντική, την ε, οικονομική μας, πρέπει όμως η βιομηχανική πολιτική να είναι ανεξάρτητη. Είναι πρωτοπόρα κίνηση αυτή εκ μέρους του κ. Λάγκια και πρέπει να την ε, ακολουθήσουμε. Επίσης, συμφωνήθηκε ο στρατηγικός στόχος να καταρτιστεί, να σχεδιαστεί αυτή η βιομηχανική πολιτική. Είμαστε πολύ περήφανοι για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες που κατά 80% βελτιώνονται κάθε χρόνο. Όμως θέλουμε να βεβαιωθούμε και για την ε, νομική, νόμιμη αγορά απασχόλησης. Έδειξε η πρόσφατη κρίση ότι είναι απαραίτητη η βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να την επιδιώξουμε. Ακόμη, η βιομηχανική πολιτική πρέπει να είναι και αποτελεσματική και έφη. οπότε Ευχαρίστω να υποβάλω τροπολογίε προ αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα καθυστερήσω με αυτά τα ζητήματα, αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Επίση, ήθελα να σταθώ στο εξή. Το θέμα τη συνεργασία. Έχουμε δει η συνεργασία να οδηγεί κάποιε φορέ σε τάσει συγχώνευση εταιριών μεταξύ διαφορετικών ε, υπήρων και στην ίδια αλυσίδα προϊόντων παραγωγή. Κάποιε φορέ υπάρχουν επιτυχημένε συνεργασίε. Αυτό συμβαίνει και από εταιρείες, με εταιρείε διαφορετικών υπηρών και σε διαφορετικού τομεί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε μια 20 ετία να ξέρουμε ότι μια αυτοκινητοβιομηχανία θα έχει και μια εταιρεία που θα ασχολείται με τι ε, τεχνολογίε επικοινωνία και πληροφορική από την Google, από τη Microsoft. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ο τομέα των νέων τεχνολογιών μπορεί να έχει μικρέ υπηρεσίε αλλού ή και αντιστρόφω. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε διορατικοί για να σχεδιάσουμε σωστά τη στρατηγική μα. Τέτοιε συγχωνεύσει βλέπουμε στι τηλεπικοινωνίε και στον ενεργειακό τομέα. Οι ενώσει εταιριών λοιπόν ε, κινούνται σε διαφορετικέ κατευθύνσει. και αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει στην, στο σχεδιασμό της βιομηχανική μας πολιτικής. Τέλος, ε, συζητήθηκε πολύ το θέμα τη χρηματοδότηση. Αλλά κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Πρέπει στην Ευρώπη να πετύχουμε να έχουμε ένα πλαίσιο φιλικό προς τις επενδύσεις για τη βιομηχανία. Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι η επενδυτική συμπεριφορά των κατώμελών δεν είναι θετική. Κάποιε φορέ χρειάζονται εξοδοτήσει και άδειε αδειών για να ανοίξει ένα εργοστάσιο. Χρειάζεται λοιπόν ένα τέτοιο περιβάλλον που να είναι φιλικό προ τι επενδύσει. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για να έχουμε μια καλή βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Τικάου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω κι εγώ κάποιες ε, παρατηρήσεις Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την πολιτική των πρώτων υλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήταν ευπρόσδεκτη μία ε, έκθεση πρωτοβουλίας προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό, αυτή η πολιτική σχετίζεται πάρα πολύ με τη βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης. Επίσης, είναι γνωστό ότι η ενεργειακή κατανάλωση θα μπορούσε να επηρεαστεί από την καλή εξέλιξη της βιομηχανίας. Αν η βιομηχανία πάρει μπρος, αυτό θα επηρεάσει και την ενεργειακή κατανάλωση. Αν αναγκαστούν να κλείσουν α, βιομηχανίες, μεγάλες εταιρείε, αυτό επηρεάζει και την ε, ενεργειακή κατανάλωση. Θα πρέπει οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις να εκμοντερνιστούν. Και αν υπάρξει εγγυημένη χρηματοδότηση προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε, να προάγουμε, να εξυγχρονίσουμε τη βιομηχανία, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη, προκειμένου να λειτουργούν με τρόπο αποδοτικό. Είναι σημαντικό να μπουν και τα συνδικάτα στη συζήτηση αυτή. Η κατάρτιση της πολιτικής της βιομηχανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδύεται με τις θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να προσελκύσουμε και τα πανεπιστήμια, την ακαδημαϊκή κοινότητα. Θα πρέπει από κοινού να αποφασίσουμε πώς θα διαμορφωθεί στο μέλλον η βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνάδελφος Γκέρεκ. Πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι χωρίς προστατευτισμό, χωρίς κρατικό προστατευτισμό, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία βιομηχανική πολιτική ούτε στις μεμονωμένες χώρες, ούτε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε μπορούμε να ικανοποιήσουμε την κοινωνία από αυτή την άποψη. Θα σας δώσω το παράδειγμα της Πολωνίας. Στην Πολωνία αυτό που συνέβη... Ε, βλέπω το χρονόμετρο. Α, προσθέσετε το χρόνο της προηγούμενης ομιλητής. Λοιπόν, ωραία. Αυτό που συνέβη στην Πολωνία είναι ότι κάποια στιγμή ανοιχτήκαμε προς την Ευρώπη και στον κόσμο, χωρίς όμως καμία αμοιβαιότητα φυσικά. Οπότε κατατροπώθηκε η πολωνική βιομηχανία από υπερεθνικές εταιρείες που είχαν πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και αγόρασαν κάποιους οικονομικούς κλάδους που ούτε τους εκαθάρισαν, ούτε τους ε, είτε οδήγησαν άλλες βιομηχανίες στην ε, εξολόθρευση. Αυτό συνέβη στην Πολωνία και αυτό φυσικά επηρέασε πολύ σοβαρά και τον προϋπολογισμό. Γιατί τέτοια έσοδα του υπολογισμού έφυγαν προς, διέρευσαν προς τις, στους προϋπολογισμούς αυτών των πολυεθνικών και προς άλλες χώρες. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα της Πολωνίας, γιατί συνέβη και σε άλλες χώρες. Η Fiat, για παράδειγμα, αγόρασε με ελάχιστα χρήματα ένα εργοστάσιο που ε, αγόρασε, που έφτιαχνε αυτοκίνητα πάντα σε μια πολωνική πόλη και μάλιστα αυτό το εργοστάσιο ήταν, ε, αντιπροσώπευε 4% του προϋπολογισμού. Είχαμε λοιπόν με αυτή τη σημαντική απώλεια στο πολωνικό ΑΕΠ όχι μόνο οικονομική, οικονομικές ζημίες αλλά και κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Χρειάζεται ο προστατευτισμός λοιπόν, ο εθνικός προστατευτισμός. Μόνο έτσι θα ξαναφτιάξουμε μια εθνική και μια ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σας ευχαριστώ, δυστυχώ εξάντλησα το χρόνο μου. Ευχαριστώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λόγο κύριος Μπέρκμαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουμε κάποιες προτάσεις που εντάσσονται στη στρατηγική του 2020. Είναι πολλές και διάφορες οι πρωτοβουλίες. Βέβαια το χρονοδιάγραμμα της έγκρισης έχει τροποποιηθεί, δεν προβλέπονται πια για για τις 27 Οκτωβρίου. Το χρονοδιάγραμμα όμως μόνο άλλαξε, αλλά όχι οι στόχοι. Οι στόχοι μας είναι να υποστηρίξουμε μια ισχυρή, ανταγωνιστική και διαφοροποιημένη βιομηχανία και βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θέλουμε η ανταγωνιστικότητα αλλά και η βιωσιμότητα να βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της ανακοίνωσης. Πρόκειται για ένα έγγραφο στρατηγικής αλλά και έγγραφο εργασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλούμε για ανταγωνιστικότητα, εννοούμε και ανταγωνιστικότητα του κόστους και των τιμών, αλλά και της καινοτομία. Και θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να διευκρινίσουμε κάτι που προκύπτει και από την έκθεση του κυρίου Λάγκε. Δεν νοείται βιωσιμότητα χωρίς ανταγωνιστικότητα και δεν νοείται ανταγωνιστικότητα χωρίς καινοτομία. Η ισορροπία στην ε, έκθεση ίσως ε, κλείνει περισσότερο προς τη βιωσιμότητα και λίγο λιγότερο ε, γέρνει προς την ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό η ισορροπία θα πρέπει να τροποποιηθεί κάπως στην έκθεση. Θα ήθελα επίσης να επικεντρωθώ σε τρία σημεία που θα αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας και ελπίζω να υπογραμμιστούν δεόντως και στο σχέδιο έκθεσης. Τρία είναι λοιπόν τα ουσιώδη σημεία. Το πρώτο είναι η σημασία ε, τη, του να προσεγγίσουμε το θέμα όχι υπό τη μορφή μονομένων βιομηχανικών κλάδων, αλλά αλυσίδων ε, είτε αξίας είτε τιμών. Γιατί κάποιες, κάποια τμήματα της αλυσίδας αυτής ε, χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους και ε, μεθεγκατίστανται. Είναι όλα σημαντικά, όλοι οι τομείς είναι σημαντικοί. Θα πρέπει να φέρουμε αντιμέτωπου στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Να μην λέμε να προωθήσουμε μόνο τους, τις πράσινες βιομηχανίες, τις φιλοπεριβαλλοντικές, εις βάρος των ε, ενεργειοβόρων, για παράδειγμα, βιομηχανικών κλάδων. Ένα άλλο σημείο είναι το εξή. Το θέμα των εθνικών βιομηχανιών που είναι απομονωμένε είναι παροχημένη έννοια. Χάρη στην ενιαία αγορά και στην ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωση δεν υπάρχουν πλέον απομονωμένε βιομηχανίε. Έχουμε πλέον διεθνεί βιομηχανίε και θα πρέπει να υιοθετήσουμε και μια διεθνή προσέγγιση και στη συγκεκριμένη μα περίπτωση ευρωπαϊκή προσέγγιση. Επίση αναφέρθηκαν και άλλε πολιτικέ όταν μιλούμε για ολοκληρωμένη προσέγγιση. Έχουμε και πολλές άλλες πολιτικές που έχουν βιομηχανική διάσταση. Περιβαλλοντική πολιτική, το θέμα της εμπορίας εκπομπών, ενεργειακή πολιτική, προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες πολιτικές λοιπόν έχουν σημαντική βιομηχανική διάσταση. Δεν είναι μόνο η βιομηχανική πολιτική. Αυτό έχει συνέπεια και για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Και αυτό το θέμα θα πρέπει να βελτιωθεί, να ενισχυθεί. Θέλουμε ευφιέστερη και πιο φιλόδοξη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και τέλος, κάτι που λείπει κάπως από την έκθεση είναι ότι μερικές φορές παρά είμαστε άτολμοι και διακριτικοί και ξεχνούμε την ισχύ που έχει η Ευρώπη. Ας μην ξεχνούμε ότι η Ευρώπη είναι μια αγορά με 500 εκατομμύρια καταναλωτές, με 200 εκατομμύρια θέσεις και 20 εκατομμύρια επιχειρηματίες. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε σε αυτή τη δύναμη που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης δεν θα πρέπει να βολευόμαστε ε, με τη συνέχιση της κατάστασης να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί οι άλλοι οι αντίπαλοι μας, οι εταίροι μας, οι ανταγωνιστές μας κινούνται με ραχθέους ρυθμούς και θα πρέπει για να είμαστε ανταγωνιστικοί μαζί τους να είμαστε και εμείς πιο φιλόδοξοι να μειώσουμε το κόστος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε- στην Ένωση και να δημιουργήσουμε την κρίσιμη μάζα των οικονομικών αλλαγών και της ανταγωνιστικότητας. Και θα πρέπει να ξεφύγουμε από την εθνική προοπτική, να υιοθετήσουμε μια πιο ευρωπαϊκή προοπτική. Όπως σας είπα, 27 Οκτωβρίου προβλέπεται η έγκριση θα συνομιλήσουμε με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για το σχέδιο της έκθεσης. Έχω πάντως την αίσθηση ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθούν την ίδια γραμμή πλεύσης. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο κλείνοντα και στον ε, εισηγητή, τον κύριο Λάγκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ενδιαφέρουσε παρατηρήσει. Δεν μπορώ φυσικά να απαντήσω λεπτομερώ στι διάφορε ερωτήσει πολλά από αυτά που αναφέρατε με απασχολούσαν και εμένα ιδιαίτερα. Κύριε Βέιμπερ, για τα θέματα χρηματοδότησης συμφωνούμε. Το θέμα επίσης της ενιαίας αγοράς, αλλά το πρόβλημα το οποίο είναι αυτό που ανέφερε και η ώρα. Ότι έχω περιορισμό και στην έκταση της έκθεσης. Πρέπει να επιλέξω λοιπόν τι θα κάνω, τι θα γράψω. Θα πρέπει όλα μαζί να καταφέρουμε να τα χωρέσω. Θα συζητήσουμε λοιπόν για τροπολογίες και χαίρομαι για το made in, την επισήμανση αυτή. Έχουμε την έκθεση Μουσκαρντίνη και την ε, Επιτροπή Εμπορίου. Το πρόβλημα όντως ε, έγκυται στα κράτη-μέλη που είναι πολύ αντίθετα. Ε, να το συζητήσουμε, πρέπει να πατήσουμε λίγο γκάζι. Χαίρομαι για τις τροπολογίες. Να σας παρακαλέσω οι τροπολογίες να εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Πραγματικά να δώσουμε μία όθηση σε στοιχεία τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη. Σας ευχαριστώ λοιπόν εκ των προτέρων και θα χαίρομαι που θα ακολουθήσουν και δικές συζητήσεις. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος, να δώσω μία συμβουλή στον κύριο Ντελάνε στον κύριο Αν θέλετε να γράψετε κι άλλα, να γράψετε βιβλίο. Σας ευχαριστώ, το ξαναλέμε στι 3, λέει ο Πρόεδρο.